Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Πρώτο σημείο στη μερίσια διάταξη, ανακοινώσεις των συντονιστών, ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών, συνεδρία των συντονιστών που έγινε χθε το απόγευμα οι συντονιστές αποφάσισαν να μην αναλάβουν μία απόφαση αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη δημιουργία ομάδας εργασίας για την τροποποίηση του άρθρου 204 του κανονισμού όσον αφορά τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Παρ' όλα αυτά, συμφωνούν με την πρόταση να δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας. Μάργαρετ στο τέλος παρεμβασίζουμε, μου παρακαλώ. Αποφάσισαν όμως οι συντονιστές να εγκρίνουν την πρόταση να ενεργοποιηθεί μάλλον να επανεργοποιηθεί μια διαδικασία για την τροποποίηση του παραρτήματος 7 του κανονισμού, όπου προβλέπεται ποια ακριβώς θα είναι ποιο θα είναι το όνομα και ποιε θα είναι οι αρμοδιότητε τη Επιτροπή Αναφορών. Θα δώσουμε λοιπόν κάποιε οδηγίε προ τη Γραμματεία, η οποία στη συνέχεια θα υποβάλει μία πρόταση και θέλουμε ουσιαστικά να επανεξετάσουμε την ονομασία της Επιτροπής μας και κυρίως να καταφέρουμε να καλύψουμε με καλύτερο τρόπο τις νέες αρμοδιότητες επιτροπής μας, όπως ακριβώς προβλέπει ο κανονισμός του Κοινοβουλίου για όλες τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Επίσης, ε, προτάθηκε και εγκρίθηκε, Μάργαρετ, σε παρακαλώ πολύ, στο τέλος παρέμβασής μου. Μπορείς να πάρεις το λόγο για όλες αυτές τις ανακοινώσεις που αφορούν στους τονιστές, στο τέλος όμως παρέμβασής μου. Προτάθηκε και εγκρίθηκε το αίτημα για μία μελέτη για μία εμβάθυνση όσον αφορά τον ε, κανονισμό και όσον αφορά τις νέες καινοτομίες που έχουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Θα ζητηθεί από τους εμπειρογνώμονες που θα επιλέξουμε να αναλύσουν με ένα πιο λεπτομερή τρόπο πώ θα μπορούσε να εφαρμοστεί με καλύτερο τρόπο ο σχετικό κανονισμό και ποιε θα είναι οι νέε αρμοδιότητε τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή και πώ θα πρέπει να λειτουργήσει στο μέλλον η επιτροπή μα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Όσον αφορά τον διορισμό των υπευθύνων εμπειρογνωμόνων, ζητήθηκε εδώ πέρα μία αναβολή της απόφασης αυτής, γιατί έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή μια καθυστέρηση για διοικητικούς λόγους και ουσιαστικά θέλουμε τα δύο αιτήματα για εκθέσεις πρωτοβουλίας που είχαν εγκριθεί στην προηγούμενη συνεδρία των συντονιστών να αναβληθούν γιατί δεν ουσιαστικά κατάφερε η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών εξετάσει το αίτημα αυτό. Επίσης εγκρίθηκε η μερίσια διάταξη με κάποιες τροποποίησεις. Η πρώτη τροποποίηση έχει να κάνει με την εισαγωγή μετά από αίτημα της κυρία Σόκεν μιας αναφοράς 1040 του 2012 και η δεύτερη τροποποίηση τη μερίσια διάταξης έχει να κάνει με την εισαγωγή σε σχέση με την έκθεση για τη Γαλλικία μιας νέας προθεσμίας για την παρουσίαση των τροπολογιών. Γιατί μετά την τελευταία συνάντηση που έλαβε χώρα δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Επομένως, το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Μπουλάντα θα έχει ως ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών την 3η Σεπτεμβρίου. Και έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε για το πρώτο τμήμα της έκθεσης αυτής, για το περιγραφικό τμήμα, τροπολογίες μόνο από όσου συμμετείχαν στην αποστολή αυτή. Για το δεύτερο τμήμα της έκθεσης αυτής μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας. Αυτό άλλωστε προβλέπεται και από, την, από τον καονισμό της Επιτροπής μας. Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Όκιν για να κάνει τις δικές παρατηρήσεις. Yeah. Uh, sorry to say... Συγγνώμη, αλλά ήταν από τις χειρότερες συναντήσεις η χθεσινή των συντονιστών στην Επιτροπή μας. Ήμουν η μόνη, εκτός από τα δύο μεγάλα κόμματα, όλα είχαν προαποφασιστεί οι... αποφάσισαν παρά την, τον έργο των αντιπροσωπιών εκ των προτέρων να μην γίνει καμία αλλαγή στους κανόνες για το όνομα κλπ. Δεν έλαβαν υπόψη το ότι δεν καταλαβαίνουν σε ορισμένε χώρες τι επιτροπή είναι αυτή και έγινε χειραγώγηση το, με βάση τους κανονισμούς. Και αυτό αφορά και την αντιπροσωπεία στη Γαλλικία όπου αποφασίστηκε ότι μόνο ο επικεφαλής έχει αρμοδιότητα, ενώ ο κανονισμός προβλέπει ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι συμμετέχοντες με πλειοψηφίες, με μειοψηφίες, έτσι γίνεται. Ενώ αποφάσι, εγώ καταψηφίστηκα γιατί ήμουν η μόνη που υπερασπίστηκα τους ε, κανονισμούς, ότι μόνο ο πρόεδρος. Οπότε πραγματικά ξεδοντιάζεται η Επιτροπή μας. Αυτό με έχει εξοργήσει και θα βρω τρόπους να το ε, κοινοποιήσω αυτό σε όλο το κοινοβούλιο γιατί είχαμε την εμπειρία από την εκλογή του διαμεσολαβητή με τις μυστικές υπογραφές παρόλο που γίνονται συστάσεις και οι συστάσεις πρέπει να κοινοποιούνται. Ενώ αυτό δεν το θέλετε και μας καταψηφίζετε εμάς. Οι μειοψηφίες πρέπει να προστατεύονται στο κοινοβούλιο. Εμείς Θέλουμε να λειτουργεί καλά η Επιτροπή. Όλα είναι σαφή, κυρία Ουκέν, διακόπτη η, πρόεδρες, η πρόεδρος. Η θέση σας είναι σαφής. Σέρε Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευτυχώς τους κανόνες δεν τους φτιάχνουν οι πολιτικές ομάδες, ούτε η πολιτική ομάδα μειοψηφία της κυρίας Χόκιν. Τους κανόνες τους φτιάχνουν οι πλειοψηφίες τις οποίες ψηφίζουν οι εκλογείς ε, στη διάρκεια των εκλογών. Στη δημοκρατία η πλειοψηφία κερδίζει όταν παίρνει τις περισσότερες ψήφους. Ως προς το θέμα της γατικίας, αυτό που σας ζητώ είναι το εξής. Χθες ελήφθη μία απόφαση με την οποία η ομάδα μου δεν συμφωνεί. Ε, ζητείται από τον κύριο Μπουλάνη η εφαρμογή του άρθρου 52 στο περιγραφικό τμήμα της έκθεσης που είχε ε, παρουσιάσει ο κύριος Μπουλάν. Προτείνω να το ψηφίσουμε αυτό, να τεθεί προς ψηφοφορία γιατί στην Ολομέλεια της Επιτροπής Αναφορών είναι αυτό που πρέπει, είναι το χώρος όπου πρέπει να ψηφιστεί κατά πόσο συμφωνούμε να εφαρμοστεί το άρθρο 52 του κανονισμού σε σχέση με την έκθεση της Γαλλικίας. Της Γαλλικίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν ακολουθήσουμε τη λογική του κυρίου Ρετουργκάης με τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες, ε, είμαστε τρία μέλη στην αντιπροσωπεία που πήγε στη Γαλλικία και η έκθεση υπευλήθη από δύο μέλη. Ε, αυτό εξετάστηκε στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι η έκθεση λοιπόν θα πρέπει να ψηφιστεί μαζί με τις τροπολογίες. Βέβαια δεν είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε σήμερα, γιατί δεν είχαμε επισήμως υποβάλει κείμενο εναλλακτικό ε, σε σχέση με το κείμενο του κυρίου Μπουλά. Δεν μας ε, διενεμήθη κείμενο μέχρι σήμερα το πρωί. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει τώρα να συζητήσουμε για το διαδικαστικό, ίσως να συζητήσουμε την έκθεση για τη Γαλλικία και να δούμε τι συνέχεια θα δοθεί. Η Αντζέλικα ε, Βίτμαν δεν είναι εδώ, αλλά δόθηκε, η Αγγέλικα Βέρτμαν ε, δεν είναι εδώ, αλλά έχει δοθεί ένα κείμενο που θεωρώ ότι είναι επίσημο και μπορεί να αποτελέσει την βάση για τη συζήτηση, διότι ε, συμφωνήθηκε από την πλειοψηφία. Μάλιστα. Συνάδελφοι, παρακαλώ μην ξανανοίξουμε ολόκληρη συζήτηση. Μόνο μια εισαγωγή με τη θέση σας και τίποτα άλλο. Ο κύριος Μπουλάμ. Διαδικαστικά μπορούμε να ψηφίσουμε πρώτα και μετά να θέσουμε τα άλλα ζητήματα γιατί αυτό ήταν ε, το αυτό που προβλέψαμε. Χρόνος, ψηφοφο... ώρα ψηφοφορίας. Να πάμε γιατί άλλοι έχουν ψηφίσουν και σε άλλες επιτροπές. Να ψηφίσουμε και μετά θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Ωραία, ωραία. Πρώτα να ψηφίσουμε και μετά να συζητήσουμε. One moment. Μισό λεπτό. La mio punto di vista. Να σας πω την άποψή μου. Εγώ διαφωνώ με την πρόταση που έγινε. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι τα μέλη της Επιτροπής μας θα πρέπει να είναι σε θέση να συμφωνήσουν αυτή τη στιγμή. Γιατί διαφορετικά εδώ πέρα ο καθένας θα εκφράσει την άποψή του, πρέπει να δούμε στη συνέχεια ποια απόφαση θα πάρουμε και πολύ γρήγορα. Εγώ νομίζω όμως το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Με αυτές τις συνεχείς αναβολές τελικά δεν καταφέρνουμε να ακούσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Συμφωνείτε πάντως μετά όσα είπε η συνάδελφος. Κανείς δεν είναι υπέρ της πρότασης που έγινε για αναβολή. Λοιπόν, ένα λεπτό και κλείνουμε όμως. Μπουλό, Μπουλάν Μέιερ και μετά κλείνουμε το σημείο αυτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με το αίτημα του Κάρλος Σιτουργκάης, δηλαδή να δούμε με ψήφο αν θα εφαρμόσουμε το άρθρο 52. Μας δώσατε 15 μέρες επιπλέον για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση. Την πρώτη εβδομάδα καμία από τις δύο συναδέλφους δεν ήταν διαθέσιμη. Τη δεύτερη εβδομάδα δόθηκε ελάχιστο χρόνος για να συναντηθώ μαζί τους. Η, κατάσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να συμφωνήσουμε για το κείμενο αυτό το οποίο υπάρχει. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει σε μια άλλη συνεδρίαση να ασχοληθούμε περισσότερο με την έκθεση αυτή. Και πραγματικά λυπάμαι που η όλη αυτή συζήτηση και η κατάσταση η οποία προέκυψε τελικά δηλητηρίασε την όλη συζήτηση. Εγώ προτείνω να εφαρμοστεί το άρθρο 52. Μέιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή αυτή άπαξ και οργανώσαμε διερευνητική επιτροπή και αποστολή Όσοι την απαρτίζουν την αποστολή είναι αυτοί που υποβάλλουν την έκθεση και αυτή είναι η δημοκρατική μέθοδος. Ο κύριος Ιτουργκάης και εγώ ε, συμμετείχαμε σε μια διερευνητική επιτροπή που μετέβη στην Αμόχωστο. Ε, τρεις ήμασταν και έγινε, ή τέσσερις και είχαμε μια συζήτηση. Δύο-δύο, δύο προς δύο, δύο και δύο. Και αποφασίσαμε λοιπόν να υποβάλουμε την έκθεση για την Αμόχωστο βάσει αυτών που είδαν οι ερευνητές όταν πήγαν επί τόπου στην Αμόχωστο. Το ίδιο θα, κριτήριο θα πρέπει να ισχύσει και με τη Γαλλικία. Και ο κανόνας της πλειοψηφία και μειοψηφία. Έτσι έχουμε δουλέψει μέχρι σήμερα. Εάν δεν συμφωνείτε, μετά ως βουλευτές παρουσιάζετε τροπολογίες. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τη θέση σας και αυτό είναι και η νόμιμη θέση. Η επίκληση του άρθρου ε, στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Μπουλάν δεν είναι σωστή. Το εξετάσαμε και είναι σφαλμένη. Και όταν αναφέρεστε το ότι υπήρξε αντιπαράθεση απόψεων, θέλω να σας πω ότι την αντιπαράθεση αυτή την οφείλουμε στη δική σας τάση και στη δική σας δράση, τη δικτατορική. Δεν θέλατε να κάνετε διάλογο είχατε την εξή θέση. Εγώ διατάζω και θα γίνει ό,τι λέω εγώ. το ουσιαστικά χειραγωγηθήκατε από το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα, προσπαθείτε να χειραγωγήσετε αυτή την Επιτροπή και προσπαθείτε να χειραγωγήσετε και τη Γραμματεία, η οποία έχει διαφυλάξει, ευτυχώ και είναι και η μόνη που έχει διαφυλάξει την αξιοπιστία τη. Γιατί υπάρχουν μέλη εδώ τα οποία δεν έχουν σωστή στάση και ειδικότερα ω προ τι ευθύνε του έναντι των πολιτών. Ευχαριστώ. Δεδομένου ότι δίστανται οι σα ζητώ να εκφράσετε μία σε σχέση με την απόφαση που ελήφθη χθε από τους τονιστές μετά από δική μου πρόταση. Επ' αυτού λοιπόν να ψηφίσουμε. Αποφασίστηκε χθε στους συντονιστές, το επαναλαμβάνω, να εργαστούμε βάσει του βασικού κειμένου που παρουσίασε ο κύριος Μπουλάντ και να παρουσιαστούν στις 3 Σεπτεμβρίου οι τροπολογίες και οι τροπολογίες αυτές μπορούν να κατατεθούν για το περιγραφικό τμήμα μόνο από τα μέλη της αντιπροσωπείας, μετά από συστάσεις μπορούν να γίνουν από τα υπόλοιπα μέλη και στη συνέχεια βέβαια μπορούν όλοι να ψηφίσουν. Ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι κατά της πρότασης αυτής. Επ' αυτού λοιπόν να ψηφίσουμε. Και αν καταψηφίσετε, αν επικρατήσει αρνητική ψήφος, τότε θα ακολουθήσουμε το πρώην άρθρο 52, όπου προβλέπεται μία εξακρίβωση του αποδεκτού της διαδικασίας αυτής, την οποία θα ήθελα πρώτα βέβαια να επαληθεύσουμε και θα απευθυνθώ γι' αυτό στις αρμόδιες αρχές. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης αυτής όπως την εξέφρασα. Το κείμενο σας δόθηκε, λέει η Πρόεδρος. Κυρία Τζανόκα, το κείμενο διενεμήθη πριν από μία εβδομάδα. Ο κύριος Λό, ο κύριος Λό με ενημέρωσε ότι ο ίδιος προχώρησε στη διαμονή του... διανομή του κειμένου αυτού. Επομένως δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από αυτού θεωρώ. Ποιος είναι υπέρ. ποιος είναι υπέρ της απόφασης που έλαβαν χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα οι συντονιστές. Ποιος είναι κατά αυτής της απόφασης. Για άλλη μια φορά, μάλιστα, λοιπόν. Η ψηφοφορία άρχεται αυτή τη στιγμή για τα όσα ανακοίνωσα ως απόφαση τελικά των συντονιστών. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Το βασικό κείμενο είναι αυτό το οποίο παρουσίασε ο κύριος Μπουλάντα. Προθεσμία η 3η Σεπτεμβρίου για την κατάθεση τροπολογιών. Οι τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν για το περιγραφικό τμήμα από όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στην αποστολή για το τμήμα των συστάσεων και για τις συμπεράσματα τροπολογίες μπορούν να υποβάλουν όλα τα μέλη της Επιτροπής και η ψηφοφορία βέβαια αφορά όλα τα μέλη της Επιτροπής. Άρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η ψηφοφορία για να μου πείτε αν είστε υπέρ της διαδικασίας αυτής ή σε περίπτωση αρνητικής απόφασής σας, αρνητικής ψήφου, ουσιαστικά είστε υπέρ του να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται από το πρώην άρθρο 52, σύμφωνα με το οποίο εγώ θα κάνω πρώτα μία επαλήθευση του παραδεκτού της πρότασης αυτής με τις αρμόδιες αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαφές τώρα για το ότι ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης αυτής παρακαλώ. Chi è favorevole a questa decisione? Υπέρ παρακαλώ πολύ της πρότασης αυτής. Τρεις υπέρ, κατά. Ο κύριος Μποστινάρου. Κυρία Πρόεδρε, το άρθρο 52 μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν δεν καταφέρουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση των συντονιστών. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Αν μέχρι το Σεπτέμβριο όχι, διακόπτη πρόεδρος. Πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το άρθρο 52, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή τη διαδικασία στα πλαίσια δηλαδή της Επιτροπής. Θα ζητήσω λοιπόν μία επιβεβαίωση για την εφαρμογή του άρθρου 52 από τη Γραμματεία για το αν μπορεί να γίνει αποδεκτό το άρθρο αυτό. Στην περίπτωση βέβαια που εγκρίνετε εσείς να εφαρμοστεί το άρθρο 52. Αν υπερψηφίσετε όμως την απόφαση των συντονιστών, τη χθεσινή, όπου αποφασίστηκε, ακριβώς επειδή είναι διδικαστικό το ζήτημα, να χρησιμοποιήσουμε και την αποστολή στη Ρουμανία την ίδια διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο σας πρότεινα χθε το βράδυ να επαναλάβουμε την διαδικασία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη διερευνητική αποστολή στη Ρουμανία. Αν τώρα αλλάξετε εσείς γνώμη και δεν θέλετε τελικά να συμφωνήσετε μετά όσο αποφασίσατε χθε το βράδυ, θα πρέπει να ψηφίσουμε και αν καταψηφίσετε την απόφαση αυτή, δηλαδή την απόφαση, τη χθεσινή απόφαση των Ιστών, τότε το ζήτημα αυτό θα περάσει στη Γραμματεία και στη συνέχεια στην Επιτροπή ΑΦΚΟ, προκειμένου να ερμηνεύσει για μας τους α, ισχύοντες κανόνες και κατά αυτόν τον τρόπο θα σταματήσουμε και την εξέταση της έκθεσης αυτής. Ξέρετε ότι στην περίπτωση αυτή θα αρχίσει μια μακρόχρονη γραφειοκρατική διαδικασία τελικά. Δική σας όμως είναι απόφαση. Θεωρώ πάντως ότι με την τροποποίηση η οποία προτάθηκε μπορείτε πραγματικά να επιτελέσετε το έργο σας ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορείτε πάντως εντελώς ελεύθερα και κατά συνείδηση να ψηφίσετε υπέρ ή κατά της πρότασής μου για μία ακόμη και τελευταία φορά ποιος είναι υπέρ της διαδικασίας την οποία προτείναμε χθε το βράδυ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των συντονιστών. Ποιος είναι υπέρ της απόφασης των συντονιστών. Μάλιστα. Βλέπω ότι η πλειοψηφία είναι κατά της διαδικασίας η οποία προτάθηκε χθε το βράδυ από τους συντονιστές. Άρα ακολουθούμε την εναλλακτική. Ποια είναι αυτή. Να ζητήσουμε μία ερμηνεία του άρθρου 52 και σταματάμε την εξέταση της έκθεσης σε αυτή τη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε στο επόμενο σημείο της μερίσια διάταξης και να σας πω όμως παράλληλα ότι όλα τα υπόλοιπα σημεία τα οποία αποφάσισαν χθε οι συντονιστές έχουν επιβεβαιωθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της μερίσια διάταξης, ψηφοφορία για την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το έτος 2012. Κύριε Σαλαβράκο, θέλετε να πάρετε το λόγο. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. με όμως τις ευκαιρίες να συγχαρώ θερμά τη νέα διαμεσολαβητή την κυρία Οράιλη για την εκλογή της και να ευχηθώ το καλύτερο στα νέα της καθήκοντα. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να ταλαιπωρήσω το σώμα. Είπα και προηγουμένως, το μόνο που έχω να πω είναι την έκφραση των θερμών συγχαρητηρίων στην κυρία Οράιλη για την εκλογή της, που πιστεύω να είναι επιτυχής και να συνεχίσει το έργο του κυρίου Διαμαντούρου, το οποίο ήταν επιτυχές. Ε, κατά λοιπά, καλώ τους συναδέλφους να υπερψηφίζουν την έκθεσή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαλαβράκο. Ας ξεκινήσουμε την ψηφοφορία για την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2012. Συμβαστική τροπολογία Α για την παράγραφο 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Γκόντσα για την παράγραφο 4. Όχι, με συγχωρείτε, λέει Πρόεδρος. 15, 16 και 17 καταπίπτουν. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 18 για την παράγραφο 6α νέο, Βασέσκου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19, Γκάμπριελ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 για την παράγραφο 6β, νέα, βασέσκου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία για την παράγραφο 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23, Χουντής Μέιερ, παράγραφος 8, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 24, Μπέκερ, για την παράγραφο 8, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25, για την παράγραφο 8α, Μπέκερ, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26, για την παράγραφο 9α, νέα, Γκάμπριελ, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Σ, για την παράγραφο 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 για την παράγραφο 12 της κυρία Ούκεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 για την παράγραφο 12 γκόντς υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 για την παράγραφο 12α, Χουντής Μέιερ. Σε δύο τμήματα, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Δεν θα ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της 31 γιατί καταπίπτει, επειδή απορρίφθηκε το πρώτο τμήμα. Περνάμε στο τρίτο τμήμα της τροπολογίας 31, υπέρ, κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία για το τρίτο τμήμα της τροπολογίας 31. Άρχεται ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται 9 υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 32 για την παράγραφο 13 του κυρίου Σαλαβράκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 για την παράγραφο 13. Βαλέζα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 για την παράγραφο 13α νέα της κυρίας Μπασέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 παράγραφος 15 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 για την παράγραφο 16 της κυρίας Κολάρσκα Μπομπίνσκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D για την παράγραφο 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε για την παράγραφο 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 για την 19 Χουντής Μέιερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 42 της κ. Μπασέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 παράγραφος 22 Κολάρσκα Μπομπίνσκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 44 και 45. Περνάμε στην 46 για την παράγραφο 22α νέα της κυρίας Γκόντς υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 για την παράγραφο 22α νέα, όκεν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 48 για την παράγραφο 22α νέα. Γκάμπριελ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 για την παράγραφο 23 της κυρίας Γκόγκς υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 για την παράγραφο 23α νέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51, παράγραφος 23β νέα, γκόνς υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 52 για την παράγραφο 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος Γα νέα, τροπολογία 1, Μπασέσκου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Όκεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7, Γκάμπριελ, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, τεχνική τροπολογία του κυρίου Σαλαβράκου, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, Γκάμπριελ, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10, Κολάρσκα Μπομπίνσκα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτει η 11, πάμε στη 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση. Άρτη ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο της έκθεσης, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Ομόφωνα, 22 υπέρ. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαλαβράκο. Terminato la seduta di, di voto. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, έκθεση ε, σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Γαλλική. Ας ακούσουμε τον επικεφαλής της αποστολής, τον κύριο Μπουλάντ αλλά όχι πάνω από τρία λεπτά, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, λιγότερο από τρία λεπτά θα κάνω. Γιατί είτε θα αποφασίσουμε μόλις ενημερωθείτε καλύτερα για το άρθρο 52 και την εφαρμογή του, είτε θα αφήσουμε το θέμα. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας πρέπει να αφουγκράζεται τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνει το πράσινο φως σε ό,τι λέει ο καθένας. Και από τη στιγμή που έχουμε μια διερευνητική αποστολή, αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που θέλω να κάνω και προσπαθώ να κάνω με την έκθεσή μου είναι να διαπιστώσω πραγματικά τα γεγονότα στην έκθεσή μου. Τόσες καταγγελίες έχουν υπάρξει από τους ε, αναφέροντες και από τις ε, τοπικές αρχές. Όλα αυτά έπρεπε να τα πάρουμε υπόψη μας. Προσπάθησα να συντάξω μια έκθεση όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική, να ακούσω τους αναφέροντες και να ε, ακούσω και την απάντηση των αρχών και των υπευθύνων. Στην έκθεσή μου, την οποία και έχετε λάβει, περιγράφονται τα γεγονότα για αυτά τα ρίας, τα δέλτα των ποταμών στη Γαλλικία. Δεν ε, περιλάβαμε όλες τις αναφορές που είχαν υποβληθεί πριν την έναρξη της αποστολής. Αναγνωρίσαμε ορισμένα γεγονότα, τα οποία υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, μόλυνση δηλαδή και ρήπανση μη επεξεργασία των λιμάτων ή των ε, υδάτων της βροχής ε, λόγω απουσίας βιολογικού καθαρισμού για το σύνολο του πληθυσμού τα μέτρα που επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που λαμβάνονται είναι όλο και πιο θετικά και αναγνωρίζονται ως τέτοια, λαμβάνονται δηλαδή μέτρα σιγά σιγά αυτό το οποίο προτείνει η τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται ότι τελικά πράγματι θα καταφέρει να ικανοποιήσει τα θεμητά ε, ε, αιτήματα και διεκδικήσεις των αναφερομένων. Νομίζω ότι είναι αρκετά αντικειμενικό αυτό που λέω. Είναι η γενικότερη εικόνα αυτή που παρουσιάζω. Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα το συζητήσουμε ξανά αυτό το θέμα όταν θα συζητήσουμε την ψήφιση της έκθεσης και τότε θα μπούμε στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Καταρχήν μια ερώτηση στη γραμματεία. Μόλις τώρα πήραμε το κείμενο. Το σχέδιο εγγράφου εργασίας με ημερομηνία 4 Ιουλίου. Μόλις τώρα το ελάβαμε. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Παρόλο που λέει 4 Ιουλίου. Δεν το έχω ξαναδεί. Και λέει και το όνομά μου, όπως βλέπετε που ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας. Δεν είμαι έτοιμη και νομίζω κανείς εκτός ίσως από τον κύριο Μπουλάν δεν είναι έτοιμος να μιλήσει για το κείμενο αυτό γιατί μου είχε δοθεί ως μέλος της αντιπροσωπείας και ένα άλλο όπως και στην Αγγέλικα Βέρτμαν από τον κύριο Μπουλάν και έπρεπε να το συζητήσουμε τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε έτοιμες. Είχαμε πει δύο η ώρα. Ξέρετε ότι εμείς απέχουμε περισσότερο από το Στρασβούργο από ότι εσείς είχατε περισσότερο χρόνο. Μας δώσετε μια καταληκτική ημερομηνία, έξι ώρα το απόγευμα και εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε στο Στρασβούργο τόσο νωρίς. Λοιπόν, Πώς εμφανίζονται, ρωτώ τη γραμματεία, όλα αυτά τα έγγραφα, γιατί σε προηγούμενες συζητήσεις ένα μόνο έγγραφο είχε ε, κατατεθεί από την ε, Αγγέλικα Βέρτμαν και μένα, είχε δοθεί στη γραμματεία. Δεν ήταν επίσημο κείμενο, σχέδιο ήταν που έδωσε ο κύριος Μπουλάν και τώρα έχουμε αυτό εδώ το κείμενο το οποίο φέρει την ημερομηνία της 4ης Ιουλίου. Σήμερα έχουμε εγώ πάντως πρώτη φορά το βλέπω στα μάτια μου. Ενημέρωσα ήδη την Επιτροπή ότι το κείμενο διενεμήθη την Παρασκευή. Εγώ έλαβα επιβεβαίωση από τη Γραμματεία ότι εστάλει με email σε όλα τα μέλη. Άρα το λάβατε την Παρασκευή. Αυτό είναι η χρονική πορεία. Ο κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σφυριλατείται μια διαδικασία την οποία δεν καταλαβαίνω, με την οποία δεν συμφωνώ και αυτό το οποίο προτείνω είναι το εξής. Το κείμενο ε, να είναι αυτό που μας προτείνει ο κύριος Μπουλάν. Τελεία και παύλα. Όχι το κείμενο της ε, αποστολής στη Γαλλικία, ε, γιατί είναι ένα κείμενο δικό σας και δύο βουλευτών. Άρα δικό σας κείμενο, όχι της αποστολής. Αυτό που ζητώ από τις δύο συναδέλφους είναι παρακαλώ παρουσιάστε ένα κείμενο. Εσείς οι δύο. Οι δυο σας, αν δεν συμφωνείτε με αυτά που λέει ο κύριος Μπουλά, παρουσιάστε ένα κείμενο. Αφού δεν έχετε ένα έγγραφο συνενετικό, παρουσιάστε δικό σας κείμενο, άλλο ο κύριος Μπουλά και τότε τουλάχιστον εγώ θα καταφέρω να λάβω υπόψη μου και να εξετάσω την άποψή σας ε, και ποια είναι η άποψή σας για την πραγματικότητα αλλά δεν συμφωνώ με το κριτήριο που παρουσιάσατε προηγουμένως. Ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, δεν υπήρχε συνεργασία πάνω στο κείμενο μεταξύ των επισήμων συμμετασχόντων. Δεν σας δόθηκε η ευκαιρία αυτή. Το κείμενο, ακόμα και αν εστάλει πριν από λίγες μέρες, το Σαββατοκύριακο, με email, παρουσιάστηκε χωρίς να έχουν προηγηθεί συζητήσεις επ' αυτού, χωρίς μια προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή λύση. Άρα το κείμενο ε, αντιπροσωπεύει μόνο τον πρόεδρο και όχι την αντιπροσωπεία. Χρειάζεται νομίζω ένα κείμενο που να αντικατοπτρίζει τις εντυπώσεις όχι μόνο του ενός συμμετασχόντος αλλά και των τριών. Μαρτίνεθ. Κυρία Πρόεδρε, αυτό το οποίο θέλω να είναι σαφές έναντι των συναδέλφων και των αναφερόντων είναι η κατάπληξή μου. 15 χρόνια είμαι μέλος σε αυτή την ε, επιτροπή και αυτό που γίνεται τώρα είναι πρωτοφανές. Έχουμε εξετάσει πάρα πολύ δύσκολες εκθέσεις, πάρα πολύ δύσκολες στη σύνταξή μου. Εγώ αυτό το οποίο θέλω είναι να εκφράσω τη στήριξή μου στην Πρόεδρο έναντι μιας ε, κατάστασης ανώμαλης θα τη χαρακτήριζα και πρωτοφανούς. Εδώ έχουμε μία αντιπροσωπεία και μπορεί μία αντιπροσωπεία να συμφωνεί ή να διαφωνεί με μία έκθεση. Δύσκολο πράγμα η έκθεση αυτό, είναι σαφές. Και μέχρι σήμερα όλοι πάντοτε κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε τα μέλη της αντιπροσωπείας να μπορέσουν να συνεργαστούν. Έχει υπάρξει όμως και στο παρελθόν τέτοια περίπτωση να έχουμε μια έκθεση για την οποία η πλειοψηφία είναι υπέρ, η μειοψηφία κατά ή το αντίστροφο. Σε αυτή την περίπτωση τότε όλοι ως μέλη επιτροπής θα το μελετήσουμε, θα δούμε τις δύο απόψεις και θα, θα επιλέξουμε ποιο θα είναι και το βασικό κείμενο που, πάνω στο οποίο θα στηριχθούμε. Με, με ταράζει αυτή η κατάσταση και με, ε, με απασχολεί ιδιαίτερως τι θα νομίζουν και οι πολίτες που παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας ε, και που είναι μέλη του ακροατηρίου. ακροατηρίου. Έχουμε μία αντιπροσωπεία τριών μελών, δύο φρονούν το α, ο ένας φρονα, φρονεί το β, ε, είναι ένας συσχετισμός δύο προς ένα. Θα υπάρξει η έκθεση που θα εκφράζει την πλειοψηφία και μπορεί αυτός που μένει μόνος του να υποβάλει τροπολογίες, παρατηρήσεις που θα εκφράζει τη διαφωνία του. Τι να κάνουμε τώρα. Ε, με καταπλήττει όμως το γεγονός ότι ε, λέγεται το εξή, ότι χθε οι συντονιστέ έφτασαν σε χ, πέτυχαν χ συμφωνία. Οι συντονιστέ όλων των πολιτικών ομάδων. Και τώρα δεν μας αρέσει ψηφίζουμε αυτό το οποίο υποτίθεται έχουν συμφωνήσει όλοι οι συντονιστές όλων των πολιτικών ομάδων και φαίνεται ότι μόνο μία πολιτική ομάδα ε, συμφωνεί με την απόφαση των συντονιστών. Άρα ε, φαίνεται οι άλλες πολιτικές ομάδες να είναι μειοψηφία έναντι της απόφασης της πλειοψηφίας των δικών τους συντονιστών. Άρα τι ζητούν, την παρέτησή τους το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε είναι να εκφράσουμε τη στήριξή μας στην Πρόεδρο και στις προτάσεις που μας υποβάλλει. Από δική μου πλευρά, αυτό που θεωρώ είναι το εξή. Ε, αν υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο που μας διανέμεται τώρα του κυρίου Μπουλάν, τον οποίο και σέβομαι απολύτω, τότε είναι προφανές ότι δεν είναι έγγραφο ε, το οποίο έχει το πράσινο φως από τα τρία μέλη της αντιπροσωπείας, αφού δύο μέλη δεν συμφωνούν με αυτή την έκθεση. Αυτό πρέπει να αναφέρεται στο έγγραφο ρητός, ότι είναι ένα έγγραφο που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ως έκθεση της αντιπροσωπείας και δεν μπορεί να φέρει τα τρία ονόματα, αφού οι δύο διαφωνούν. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω με το έγγραφο του κυρίου Μπουλάν ή με το έγγραφο των άλλων δύο συναδέλφων, αλλά είναι ε, παραγραφή, πλαστογράφηση της πραγματικότητας να λέμε ότι το έγγραφο αυτό εκφράζει την αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω. Είχα μια συζήτηση όπου προείδρευα για ιατρικά θέματα. Εμείς προσπαθήσαμε πολύ να βρούμε συμβιβαστική λύση που σε κάποιες λεπτομέρειες απέτυχε. Δεν είναι καλή διαδικασία πιστεύω αυτή. Η συνάδελφος Τατιάνα και εγώ πιστεύουμε ότι οι αντιλήψεις μας μετά από οι συζητήσεις, αυτά που ε, είδαμε παρουσιάζονται αντικειμενικά, είναι αντικειμενικές. Πρώτα στην έκθεση θα πρέπει να αναφέρονται αυτά που είδαμε και να παρουσιάζονται τα πράγματα όπως μας παρουσιάστηκαν εκεί. Δεν χωρούν ερμηνείες εκεί και αιτήματα αυτά, θα τα επεξεργαστούμε στις συστάσεις και παρακαλώ τους συναδέλφους που πιστεύουν ότι η Τατιάνα και εγώ δεν είμαστε αρκετά συμβιβαστικές να λάβουν υπόψη αυτό το αντικειμενικό στοιχείο γιατί καθήκον μας ε, ημών των πολιτικών είναι να εφιστούμε την προσοχή στα αντικειμενικά στοιχεία. Και αν μας ρωτήσουν για τη γνώμη μας, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά δεν συζητείτε αυτό. Είμαστε Επιτροπή Αναφορών και την άποψή μου μπορώ να την επαναλάβω εδώ. Ως Επιτροπή Αναφορών πρέπει να ασχολούμεθα με τις αναφορές και όχι την κομματική πολιτική. Εγώ δεν θα επέτρεπα ποτέ στο κόμμα μου να με επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να ε, είναι σε βάρος των αναφερόντων. Παρακαλώ λοιπόν να γίνει αποδεκτό ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία. Ευχαριστώ. Μιράντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μεταξύ όλων αυτών των οπισθοχωρήσεων και πισωγυρισμάτων και ακροβασιών έχουν περάσει πέντε μήνες διαπραγματεύσεων. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες πολιτών. Συνεχώς στέλνουν mail σε βουλευτές όπως εμείς που τους έχουμε αφουγκραστεί και είμαστε δίπλα τους από την αρχή. Στο γραφείο μας φτάνουν αναρρύθμιτα σχόλια αναφερόντων που μας ρωτούν τι γίνεται με αυτή την έκθεση τέλος πάντων, τι γίνεται με την αναφορά μας. Πνιγόμαστε σε μια διοικητική διαδικασία, σε διάφορες ερμηνείες περί του κανονισμού και δεν εξετάζουμε την ουσία του προβλήματος, που είναι να λύσουμε το πρόβλημα της μόλυνσης, να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα, να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι έχει μια αξία και μια χρησιμότητα αυτή η Επιτροπή. Κύριε Βουλά, η αξιοπιστία σας είναι καταβαραθρωμένη αυτή τη στιγμή. Πήγατε στη Γαλλικία, θελήσατε να είστε αντικειμενικός, είδατε τα γεγονότα και τώρα η αξιοπιστία σας έχει υποστεί ένα πλήγμα ανεπανόρθωτο. Δηλαδή κανείς δεν θα σας ακούσει πλέον με τέτοια χαμηλή αξιοπιστία. Ποια θα είναι η εικόνα του κυρίου Μπουλάν και το λέω και σας, σέβω, σας σέβομαι απολύτως, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η πολιτική σας εικόνα όταν δεν φανήκατε αντάξιος των προσδοκιών των πολιτών και ξεπουληθήκατε στα συμφέροντα τα διάφορα με έλλειψη διαφάνειας. Και σας το λέω ειλικρινά, επιμένω και έναντι της γραμματείας. Όλες οι ελπίδες που είχαν αναποθέσει στο πρόσωπό σας χιλιάδες πολίτες έχουν αυτή τη στιγμή καταβαραθρωθεί γιατί κρύβεστε όλοι πίσω από τη γραφειοκρατική διαδικασία για να μην υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των πολιτών. Εσείς, κυρία Πρόεδρε, πράγματι υπερασπίζεστε τα, τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε πάνω σε ε, μια έκθεση την οποία περιμένουν πάρα πολλοί αναφέροντες από το 1999 το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε μια έκθεση η οποία λέει ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά, βαίνουν καλώς και να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η έλλειψη διαφάνειας η οποία επικρατεί. Άλλωστε η αντιπροσωπεία αποτελείται από τρία επίσημα μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και ελπίζω ότι θα με υποστηρίξετε και τους επόμενους μήνες για να καταφέρουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι υπέρ των πολιτών. Ο συνάδελφος Γιάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Λυπάμαι πάρα πολύ που πάλι μπήκαμε στη συζήτηση για τα διαδικαστικά. Εδώ δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την έκθεση. Θα γίνει σε δύο μέρη. Το δεύτερο μέρος είναι τα συμπεράσματα που θα ψηφιστούν εδώ στην Επιτροπή και όλοι θα κάνουν προτάσεις και τροπολογίες. Τώρα είναι το πρώτο κομμάτι, το περιγραφικό όπως λέμε και συμφωνήσαμε ότι αυτό πρέπει να ε, στηρίζεται στην ομοφωνία. Άκουσε Μάργαρετ τι λέω γιατί αυτό είναι η προστασία των μειοψηφιών. Όλοι, όλοι, αυτό σημαίνει ομοφωνία. Όλοι πρέπει να συμφωνήσουν και δεν μπορεί να ε, επικρίνεται η γραμματεία η οποία μας βοηθάει. Βοηθητικά δρά. Υπάρχουν τρεις βουλευτές εδώ που πρέπει να συμφωνήσουν εδώ ε, δεν συμφωνείτε εν προκειμένου, δεν θα ανακατευτώ να ρωτήσω το γιατί, πάντως δεν υπάρχει συμφωνία. Και αυτό πρέπει να το προβλέψουμε. Γιατί εδώ να, δεν συμβαίνει, δεν υπάρχει ομοφωνία. Το συζητήσαμε και χθε και σήμερα και αύριο θα το ξανασυζητήσουμε. Πρέπει να προβλέψουμε τι γίνεται όταν δεν υπάρχει ομόφωνη θέση. Είπαμε, αυτό το περιγραφικό κομμάτι που είναι τα στοιχεία, αυτά που πάνε και βλέπουν και τα καταγράφουν οι συμμετέχοντες, αυτά βλέπουμε ότι δεν μπορούν να τα δώσουν για να περάσουν από την Επιτροπή, γιατί δεν συμφωνούν οι συμμετασχόντες. Η ε, ομοφωνία λοιπόν στο περιγραφικό σημαίνει 100% ανεξάρτητα από το ποιο συμμετέχει. Τέλος, ελπίζω ότι το συμπέρασμα από εδώ θα είναι ότι ε, ε, ε, το συμπέρασμα να μην είναι να κάνουμε με ένα μέλος διερευνητικές αποστολές, αυτό θα ήταν ανόητο. Θα πρέπει πάντως να τα συζητούμε όλα αυτά και να υπάρχει ομοφωνία. Φταίει και ο επικεφαλής, πάντως οι διερευνητικές αποστολές συνήθως θα πρέπει να επιταχύνουν τη διαδικασία των αναφορών. Αυτά που γίνονται εδώ δείχνουν ότι συμβαίνει το αντίθετο. Συμφωνήστε, βρείτε μια, ε, έναν κοινό τόπο, αλλά όπως είναι το πρόβλημα εδώ πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει ομοφωνία. Γι' αυτό είχαμε και τρεις συμμετέχοντες με την προοπτική ότι θα συμφωνούσαν. Κύριο Σάντσεφ, ευχαριστώ πολύ. Ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα είναι να αποφύγουμε τους αρνητικούς χαρακτηρισμούς και τις επικρίσεις. Καλό είναι να αναλάβουμε όλη την ευθύνη μας. Η αντιπροσωπεία μετέβη στη Γαλλικία τον Φεβρουάριο και το φυσιολογικό θα ήταν αυτή τη στιγμή να είχαμε ήδη εγκρίνει ένα τελικό ψήφισμα. Ενώ δεν έχει συμβεί αυτό και συνεχίζουμε να συζητούμε το κατά πόσο η έκθεση αυτή εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει τα μέλη της ε, αποστολής ή όχι. Περιπλέκουμε το εύκολο και δεν ασχολούμαστε με την ουσία από διαδικαστικής πλευράς, εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Εμείς θέλουμε να βρούμε μια λογική λύση. Θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο ευέλικτοι. Θα συνεργαστούμε. Το βασικό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε είναι το εξής. Η αντιπροσωπεία έλαβε χώρα χωρίς κανένα πρόβλημα μεταξύ των συνιστοσών της. Το τι έχει γίνει το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι πολύ περίπλοκο να υπάρξει συνενετικό πόρισμα και τα υπόλοιπα είναι επίσης σαφή αυτά που πρέπει να κάνουμε. Να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στις ισπανικές αρχές, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αυτόνομης κοινότητας και της εθνικής κυβέρνησης ότι πρέπει να εφαρμόσουν το ευρωπαϊκό, το κοινοτικό δίκαιο. Και δεν μπορούν να μην το εφαρμόζουν και από την άλλη ε, να αξιοποιούν τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά. Θα πρέπει να στηριχθούν στα ευρωπαϊκά ταμεία για να μπορέσουν να εφαρμόσουν το κοινοτικό δίκαιο. Ο κύριος Μίλε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε ένα μεγάλο μπέρδεμα εδώ, αλλά ξέρουμε και από πού προέκυψε. Ένα έγγραφο κυκλοφόρησε από την γραμματεία πριν από δύο μήνες χωρίς την έγκριση του Προέδρου. Πριν από ένα μήνα δύο μέλη της αντιπροσωπείας κυκλοφόρησαν επίσης έγγραφο χωρίς την έγκριση του Προέδρου της αντιπροσωπείας και τώρα παραπονιούνται που ο ίδιος ο Πρόεδρος της αντιπροσωπείας κυκλοφορεί το δικό του έγγραφο. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κατά τη γνώμη μου όχι. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερον, Ξέρω ότι ο κύριος Μπουλά έχει κάνει πολλές προσπάθειες να πετύχει συνένεση και έχει κάνει πολλές προσπάθειες να μιλήσει με τις δύο κυρίες. Θεωρώ ότι ήταν δύσκολη η συνένεση πριν από 15 ημέρες. Όταν εσείς τα συντονίζατε αυτά κυρία Πρόεδρε, τώρα η συνένεση είναι αδύνατη να μελετήσετε την εφαρμογή του άρθρου 52. Και θεωρώ ότι αυτό που θέλουμε είναι μια αντικειμενική έκθεση θετική για τις αρχές, θετική για τη Γαλλικία, για να υπάρχουν ευρωπαϊκά ταμεία, ισορροπημένη έκθεση θετική για τους πολίτες που θέλουν να είναι καθαρά τα δέλτα και όλα τα νερά των ποταμών. Ο κύριος Μπουλάν είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας και ε, το Και αυτό το οποίο ε, θέλει να κάνει είναι να βρει συνένεση. Όλοι κυκλοφόρησαν έγγραφα εκτό από τον ίδιο. Προσπάθησε να βρει άλλη λύση, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και είναι λογικό που κυκλοφόρησε το δικό του προχθέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για να απαντήσουν έχουν ζητήσει το λόγο, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε πάρα πολύ γιατί έχουμε αναφορέ που πρέπει να συζητήσουμε. Επομένω, μην μιλήσετε για πάνω από ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Τζανόκα, Μπουλάν και Όκεν. Αυτοί οι τρει κλείνουμε το σημείο αυτό. Κύριε Τζανόκα, έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. Επί του εγγράφου. Καταρχήν, βλέπετε ότι το πρώτο μέρος μαζί με τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις είναι στα αγγλικά. Και αυτό ήταν το κείμενο που είχαμε να συζητήσουμε την περασμένη ε, Δευτέρα με τον κύριο Μπουλάνη και την Παρασκευή κυκλοφόρησε κάτι καινούριο που περιλαμβάνει συστάσεις γραμμένες στα γαλλικά. που και όλο το Σαββατοκύριακο να δουλεύαμε με την κυρία Βέρτμαν δεν θα τις επεξεργαζόμαστε. Εγώ δεν είμαι έτοιμη να συζητήσω τις συστάσεις, αν και διαβάζω γαλλικά. Η συνάδελφος δεν δυσκολεύεται. Τώρα, για τα συμπεράσματα. Στοχεύαμε στη συνένεση, αλλά αξιότιμα μέλη της αντιπροσωπείας. Αν πάρουμε το κείμενο αυτό που παρουσίασε ο κύριος Μπουλάν, αν το δεχτούμε αυτό, δεν είχε νόημα να πάμε στη Γαλλικία, γιατί εδώ απορρίπτονται 100% όλα Όλες οι ανησυχίες για την εγκατάσταση στο Ριγκανόσα λέει μόνο ότι ε, κατασκευάστηκε με βάση το ισπανικό δίκαιο και δεν λέει ότι στα 50 μέτρα έχει σπίτια. Δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση όταν η προσέγγιση του Προέδρου είναι απορριπτική όλων των μελημάτων των αναφερόντων. Ενώ η δική μας η προσέγγιση που υποστηρίζει τους αναφέροντες ε, ήταν ιδεολογικά και πολιτικά διαφορετική να κάνετε, να καταθέσετε τροπολογίες. Η κυρία Άουκεν, να ζητήσουμε ε, από την νομική υπηρεσία να κάνει ερμηνεία των κανόνων που διέπουν τις αντιπροσωπείες. Γιατί κάποιος εδώ φαίνεται ότι πιστεύει ότι ε, υπερέχει ο πρόεδρος και μπορεί να αποφασίζει αν δεν υπάρχει συμφωνία. Ενώ οι κανονισμοί δεν το λένε αυτό. Και να ε, ακολουθήσουμε την πρόταση Μαρτίνες που μιλάει για πλειοψηφία-μειοψηφία. Δεν αναφέρεται τίποτα για τον επικεφαλής ακόμα και αν οι άλλοι ε, είναι διχασμένοι. Καταρτίζεται από τους συμμετέχοντες τα κείμενα. Αν Για να μην ε, συνεχίσουμε να διαπληκτιζόμεθα, να μας πει η νομική υπηρεσία πώς ερμηνεύεται ο κανόνας θα, ο, θα τα αποφασίζει όλα ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας ή θα συμμετέχουν οι συμμετασχόντες. Να ζητήσουμε αυτό και να σταματήσουμε τη συζήτηση, γιατί εγώ δεν δέχομαι πολιτική ερμηνεία του κανόνα 202. Ο κύριος Μπουλάν, τελευταίος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω πολύ καλά το ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι θέλουν αυτή τη στιγμή να προωθήσουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων πολιτών από συγκεκριμένε περιφέρειες. Θα πρέπει όμως παρόλα αυτά να συνειδητοποιούμε ότι θέλουμε να ακούμε πάντα τους Ευρωπαίους πολίτες στα πλαίσια των αντιπροσωπιών αυτών και των επισκέψεων. Αυτό ακριβώς κάναμε και του δώσαμε και τη δυνατότητα επίσης να απαντήσουν και να φέρουμε ιδίω στις Ισπανικές Αρχές της Γαλλικίας. Η απάντηση που δόθηκε από τις Ισπανικές Αρχές ε, αξιολογήθηκε σε μια δεύτερη φάση και συζητήθηκε από την αντιπροσωπεία μας, ε, την τριμελή αυτή. Δεν μπορούμε όμως στα πλαίσια της τριμελούς αυτής αντιπροσωπείας να αντιταχθούμε σε κάποιες αποφάσεις που έχει πάρει η Ισπανική δικαιοσύνη. Να λέμε δηλαδή ότι ε, υπήρξε κακή μεταχείριση των δημοσίων χρημάτων. Δεν μπορούμε να, κάνουμε, να καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα τέτοια. Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να δούμε ποια είναι η ευθύνη μας. Εγώ αυτό ακριβώς ε, θέλω να λάβω, την ευθύνη που έχω ως επικεφαλής αντιπροσωπείας, να δώσω δηλαδή τον απαραίτητο χρόνο σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και να καταφέρω να τον δυνατόν πιο αντικειμενικός γίνεται. Όταν αποφασίσαμε εν τέλει να μην λάβουμε υπόψη μας κάποιες αναφορές, τότε εγώ είπα ότι δεν μπορούσα να αντιταχθώ στη γενική απόφαση που είχε πάρει η ομάδα μας. Διακόπτη πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπάθησα πραγματικά να καταλήξω μια συνένεση. Τον κύριο Μαρτίνες δεν τον διακόψει Τον μίλησε 4,5 λεπτά τη γιατρία. Θα ήθελα απλώς να σας πω, μα ήταν ο πρώτο γύρο ομιλιών. Είναι ο δεύτερος γύρος και σας δίνω μόνο ένα λεπτό, σας είπα. Αναζητήθηκε συνένεση, αυτό ήθελα να σας πω και λυπάμαι πραγματικά που οι συνάδελφοί μου δεν βρήκαν τον απαραίτητο χρόνο, δεν αφιέρωσαν τον απαραίτητο χρόνο για να βρεθεί αυτό, αυτή η συνενετική προσέγγιση. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστώ όλους. Κύριε Μαρτίνε, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μία παρατήρηση και βλέπω ότι για πρώτη φορά συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση που έχει κάνει η κυρία Όκεν και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πραγματικά άχρηστη όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται η Επιτροπή μας αποφάσισε να, να απευθυνθεί στη νομική υπηρεσία προκειμένου να ερμηνευθούν οι κανόνες, οι διαδικαστικοί και κατά αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε. Σήμερα το πρωί επέτρεψα να γίνει μια συζήτηση ακριβώς επειδή δεν θέλω εγώ να παρακάμψω τις δημοκρατικές διαδικασίες, πάντως θα πρέπει να ασχοληθούμε πραγματικά με την ουσία. Και πρέπει να σας πω ότι με τη δική μου την πρόταση, την οποία δεν αποδέχθηκε η Επιτροπή μας και το δέχομαι αυτό βέβαια, η δική μου πάντως η πρόταση είχε να κάνει με μία συσσωρευμένη εμπειρία που έχουμε από το παρελθόν. Ενδεχομένως να έχει γίνει κάποιο διοικητικό λάθος και το ότι υπήρχε όντως το πρόβλημα αυτό με την έκθεση του κυρίου Μπουλάντη, η οποία όμως νομίζω ότι έφτασε σε όλες τις αντιπροσωπείες και σε κάθε αντιπροσωπεία που είχαμε κάνει στο παρελθόν, σε κάθε επίσκεψη που είχαμε κάνει στο παρελθόν, είτε πρόκειται για την Ιταλία, είτε πρόκειται για την Πολωνία, πάντα έχουμε ένα κείμενο το οποίο καταδεικνύει το όνομα του εισηγητή. Αυτό κάνουμε και στην περίπτωση αυτή μπορείτε πραγματικά να επαληθεύσετε όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία έχουμε στην ιστοσελίδα μα. Πάντα ο επικεφαλή αντιπροσωπεία θεωρείται και ο εισηγητή, ο οποίο υποβάλλει το βασικό κείμενο. Εγώ με τη δική μου την πρόταση ήθελα να σα κάνω να συμμετέχετε όλοι. Γιατί ουσιαστικά όλοι θα μπορούσαν και οι συνάδελφοι δηλαδή του κυρίου Μπουλάντ να υποβάλουν ένα εναλλακτικό κείμενο. Ανταυτού Έχουμε μπλοκάρει την όλη διαδικασία ακριβώ επειδή δεν θέλατε να δεχθείτε την πρόταση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να αναμένουμε τώρα την πρόταση της νομικής υπηρεσίας. Ξέρετε ότι είχαμε καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες στο παρελθόν, όπως στην περίπτωση της επίσκεψης στη Ρουμανία. Χάνουμε αυτή τη στιγμή όμως πάρα πολύ χρόνο και πραγματικά τίθεται να αμφιβόλω η ίδια εξοπιστία της Επιτροπής μας. Μία αποστολή πραγματικά πρέπει να αποτελεί προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να βοηθά επιπλέον τους πολίτες και να μην μπλοκάρει την απάντηση αυτή την οποία τόσο καιρό περιμένουν οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν την ε, αδράνεια των τοπικών αρχών. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι στην αδράνεια των τοπικών αρχών προσθέτουμε τη δική μας την αδράνεια και αυτό δεν μας τιμά καθόλου. Έτσι λοιπόν, όπως αποφασίστηκε στην αρχή της σημερινή μας συνεδρίασης, θα ζητήσουμε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και θα σας ενημερώσω στη συνέχεια για την απόφασή τους. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, αναφορά 938 του 2012, την οποία επέβαλε η Ματίλντε Φοντέν, Ισπανικής Ιθαγένειας, η οποία είναι παρούσα. και της δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Με συγχωρείτε, πρόκειται για έναν κύριο. Σα το συγγνώμη, λέει η πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ερχόμαστε από το Δέλτα του Εύρου και μιλούμε εξ ονόματος της πλατφόρμας υπεράσπισης του Δέλτα του Εύρου. Είμαστε μια συλλογικότητα πολιτών. Επί δεκαετίες αγωνιζόμαστε ε, ώστε να υπάρξει Δέλτα στις εκβολές ε, του ποταμού Εύρου το οποίο πράγματι υποστηρίζει και προστατεύει πάρα πολλά είδη ζωικά και φυτικά. 100.000 κάτοικοι είναι εκεί. Όλες οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το Δέλτα του Εύρου υποχωρεί αυτή τη στιγμή εισβάλλει η θάλασσα, τα αλμυρά ύδατα και όλα αυτά έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις συνθήκες υγιεινής ε, των ατόμων αλλά και στην επιβίωση του οικοσυστήματος και στη σταθερότητα του Δέλτα. Θέλουμε να μειώσουμε τις κήτες των ποταμών που φτάνουν σε αυτές τις εκβολές. Ε, ε, αντλούνται υπερβολικά πολύ οι υδάτινοι πόροι και οι οποίοι σιγά σιγά στερεύουν ενώ η αλλαγή στις κλιματικές συνθήκες είναι όλο και πιο εμφανής. Το Δέλτα του Εύρου είναι ένα οικοσύστημα που έχει μελετηθεί κατά κόρον. Πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες στην Ισπανία και σε όλο τον κόσμο έχουν ταχθεί υπέρ της προστασίας αυτού. Θα θυμάστε την υψηλή, την έντονη κοινωνική, πολιτική και επιστημονική κινητοποίηση στην Ισπανία με το υδρολογικό σχέδιο το εθνικό του 2001. Το, ο βασικός σκοπός του, αυτού του σχεδίου ήταν η εκτροπή του Εύρου, ε, του ποταμού αυτού, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της εκτροπής στο δέλτα του Εύρου. Θέλουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να σημάνουν αυτό το καμπανάκι στην Αγερμού, γιατί αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, υπερεκμετάλλευσης του ποταμού Εύρου θα έχει τεράστιο ε, περιβαλλοντικό αντίκτυπο και θα καταστρέψει τελικά το δέλτα του. Η Ευρώπη δεν θέλησε να υιοθετήσει αυτή την ευθύνη. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θεωρούν ότι η περιβαλλοντική πολιτική είναι ε, μία από τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τη χαρακτηρίζουν αυτή καθεαυτή, η πιο προφανής αξία μάλιστα. Εμείς ως πολίτες και ως συλλογικότητα συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θεωρήσαμε ότι η οδηγία πλαίσιο για τα νερά θα μας προσέφερε χρήσιμα εργαλεία για να ε, σώσουμε όλα αυτά τα πολύ πολύτιμα οικοσυστήματα που διαβιούν καθόλου το, τη διαδρομή του Εύρου αλλά και στο Δέλτα του κυρίως. Φαίνεται όμως ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται δυστυχώς. Έχουν υπάρξει νέα υδρολογικά σχέδια προσαρμοσμένα στην εθνική νομοθεσία και το Ισπανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω της Συνομοσπονδίας της Γεωγραφικής για το Εύρο καθυστέρησε πέντε ολόκληρα χρόνια μέχρι ότου να συντάξει υδρολογικό σχέδιο. Και όταν το συνέταξε, ποιο συμπέρασμα έβγαλε ότι από 750.000 θα πάμε σε πάνω από 1,5 ε, εκατομμύριο εκτάρια επιπρόσθετα που θα αρδεύονται από ε, τον ποταμό Εύρο. 14.000 ε, εκατοστό κυβικά, κυβικά εκατοστά με συγχωρείτε, νερού θα αντλούνται ε, για λόγους άρδευσης, ακόμα περισσότερο. Το υδρολογικό ε, σχέδιο προβλέπει κατασκευή 35 νέων φραγμάτων και έχει και προοπτική για άλλα 44. Δηλαδή, η περιβαλλοντική κήτη που είναι απαραίτητη για να διατηρήσει τον, το Δέλτα είναι 3.000 μόνο κυβικά εκατοστά νερού. Άπαξ και ε, ε, πάρουμε το 1.400.000 που χρειαζόμαστε για τα νέα εκτάρια που θα πρέπει να αρδρευτούν, αυτά τα 3.000 κυβικά εκατοστά είναι αυτά που μένουν και γι' αυτό τα βάλαν σε αυτό το σχέδιο. Ελάχιστα κατά τη γνώμη μας. Σύμφωνα με το σχέδιο, το 70% ε, των υδάτων είναι σε καλή κατάσταση στον ποταμό Εύρο, παρόλο που περιέργως αναγνωρίζουν ότι αν μόνο τις 314 από τις 600 τόσο. Δηλαδή πώς ξέρουν ότι το 70% είναι σε καλή κατάσταση όταν έχουν μελετήσει δειγματολεπτικά το 50% μόνο. Το υδρολογικό σχέδιο επίσης δεν αξιοποιεί κάποιους από τους πιο βασικούς δείκτες, όπως είναι τα ψάρια, για παράδειγμα. Το χειρότερο με αυτό το υδρολογικό σχέδιο είναι το εξής δεν περιλαμβάνει καμία από, κανέναν από τους 14 όγκους υδάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το υδρολογικό σχέδιο του Ισπανικού ε, Υπουργείου Περιβάλλοντος, το 100% του Δέλτα του Εύρου δεν είναι ούτε σε καλή ούτε σε κακή κατάσταση. Γιατί, γιατί δεν το μελέτησαν καθόλου, αποσιάζει. Στην πράξη πώς μεταφράζεται αυτό, ότι δηλαδή το τελικό Το τελικό κομμάτι του ποταμού Εύρου, το δέλτα του, θα έχει νερά. Η κήτη του ποταμού θα είναι μικρότερη από 100 κυβικά ε, μέτρα το δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια 10 από τους 12 μήνες το χρόνο. Είναι ελάχιστο αυτό και όλο το υπόλοιπο δηλαδή θα πλημμυρίζεται από αλμυρά ύδατα της θάλασσας, κάτι το οποίο θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Με τα 35 νέα φράγματα και με τη διατήρηση των προσδοκιών για 44 νέα φράγματα δεν λαμβάνεται κανένα συγκεκριμένο μέτρο που ε, να ε, αντισταθμίζει την ανάκτηση του κόστους. Δηλαδή θα δορηθούν υποδομές στους χρήστες των αρδεύσεων χωρίς να γνωρίζουμε ποιος θα πληρώσει. Δεν έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου στα φράγματα αυτά ποιος, ε, θα είναι ο αντίκτυπος στα ειζήματα, ούτω ώστε να μην υπάρξει τόσο έντονη διάβρωση. Οι, οι Ισπανικές αρχές δεν επέτρεψαν καμία ε, κοινωνική συζήτηση. Τα τελευταία 20-30 χρόνια δεν έγινε καμία τεχνική ή πολιτική συζήτηση για τις προτάσεις, για τις κίτες του ποταμού, για τις αρδεύσεις. Ε, η μόνη τεχνική συζήτηση που κάναμε ήταν το 2003 κατόπιν ε, παρακίνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ισπανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος ποτέ δεν θέλησε να συζητήσει τα τεχνικά στοιχεία. Αυτό που υιοθέτησε ως κανόνα ήταν η διακριτικότητα και η όσο το μεγαλύτερη απόσταση από τη διαφάνεια. Γνωρίζουμε πόσες δυσκολίες αντιμετωπίσατε για να μας επιτρέψετε να είμαστε εδώ παρόντες σε αυτή την Επιτροπή και σας ευγνωμονούμε πραγματικά. Ερχόμαστε από μια πολύ μικρή περιοχή. Υπερασπιζόμαστε όμως ένα δίκαιο σκοπό που ξεπερνάει τα στενά όρια του χωριού, της κοινότητας, της επαρχίας ή της χώρας μας. Μιλούμε για μια, ένα κοινό κτήμα της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς στη Μεσόγειο, σε όλο τον κόσμο που χαίρει ε, τις προστασίας της UNESCO. UNESCO επίσης. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή και τίθεται ε, και διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία όλων μας αλλά και η επιβίωση πραγματικά ε, του Δέλτα αυτού. Ζητούμε από την Επιτροπή να μελετήσει τη διαδικασία εναρμόνισης, ενσωμάτωσης ε, στην ε, νομοθεσία του υδρολογικού ε, σχεδίου για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Εύρου και προσπα... θέλουμε να ε, προτείνετε τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα ώστε να μην εγκριθεί τελικά ένα υδρολογικό σχέδιο το οποίο στην πράξη θα σημάνει την πιο εσχρή ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα οδηγήσει τελικά στην εξαφάνιση του Δέλτα του ποταμού Εύρου, υποτίθεται εξ ονόματος της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Δίνουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Τζιοβάνι Βαλέρα. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους υπόλοιπους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε και ευχαριστώ τον αναφέροντα που ήρθε από την Ισπανία να μας τα πει όλα αυτά. Ε, θέλουμε και εμείς να πούμε δύο λόγια σήμερα. Όπως γνωρίζει ο αναφέρον, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα έχει κάποια διαδικασία. Προβλέπει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τα, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μετά από διαδικασία διαβουλεύσεων τώρα σχεδιάζεται η εγκατάσταση. Δεν είναι κάτι που αξιολογείται σε αυτό το στάδιο με βάση την ίδια την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Ε, θα λειτουργήσει και θα υπάρξει η ακθεση των Κομισιόν. Βέβαια, ο αναφέρον παρακολουθεί τα άλλα προαπαιτούμενα της ε, Οδηγία ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις για τις εγκαταστάσεις. Τώρα αναφέρονται κάποια προβλήματα και υποθέτω ότι θα έχουν κοινοποιηθεί και στις ισπανικές αρχές τα προβλήματα αυτά. Εμείς παρακολουθούμε τη διαδικασία από κοντά ώστε η Ισπανία να δώσει τα σχέδια και μάλιστα τους πήγαμε και στα δικαστήρια και κερδίσαμε την υπόθεση ευτυχώς. Κάναμε ό,τι είναι δυνατόν για να τα ε, καταφέρουμε αυτά και η νομική υπηρεσία μας εργάζεται ε, για να βοηθήσει να υιοθετηθούν τα προγράμματα και μετά σιγά σιγά θα αξιολογηθούν τα ε, προγράμματα αυτά. Αυτό θα πάρει χρόνο και θα δεχθούμε και σχόλια για τα καινούργια τις καινούργιες εγκαταστάσεις ε, όταν θα εγκριθούν. Επίσης είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας εδώ ότι όταν τα σχέδια εγκριθούν θα πρέπει να εξεταστούν, όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε σχέδια επισχεδίων τώρα σχέδιο, πάνω στο σχέδιο. Να με διορθώσει ο αναφέρον, αλλά νομίζω ότι σήμερα, ότι στις 4 Ιουλίου, το, σχέδιο, το πρώτο σχέδιο δόθηκε στο αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά πρέπει να πάει στο Εθνικό Συμβούλιο, να περάσει από την κυβέρνηση, δηλαδή ακόμα μέλουν πολλά να γίνουν. Και κάθε φορά πρέπει να, υπό, να λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια για τη λεκάνη του ποταμού. Ελπίζομαι ότι κάποια στιγμή θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο. Η Ισπανία μας έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το παρακολουθούμε. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, γιατί ακόμα και αν ε, προσφέγουμε στο δικαστήριο κατά της Ισπανίας για τα σχέδια, αν δεν ε, συμμορφωθεί θα περάσουν άλλα δύο χρόνια. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε προσπάθειες για να έρθει ένα σχέδιο και να δούμε αν συνάδει με την οδηγία. Όπως κάναμε και με άλλα κράτη-μέλη που έδωσαν σχέδια. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων πριν να υποβληθούν τα σχέδια να ε, προχωρήσουμε σε κατά μέτρα εξαναγκασμού της ε, χώρας μέλους. Ευχαριστώ που ήρθατε. Νομίζω ότι κάνετε μέχρι τώρα τη δουλειά σας πάρα πολύ καλά γιατί κάνετε αυτό που προβλέπει η οδηγία να υποβληθούν τα σχόλια και τώρα η Ισπανία θα πρέπει να ανταποκριθεί. Ε, πρέπει να δούμε όμως τα τελικά σχέδια και θα ε, δεχθούμε ευχαρίστως τα σχόλιά σας όταν θα μας κοινοποιηθεί το τελικό σχέδιο όπως, ε, δηλαδή θα ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθήθηκε και σε άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε τον γύρο παρεμβάσεων. Η κυρία Λόπεθ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, Όσον αφορά στην ε, αναφορά της κυρίας Ματίλντε Φόντς για την πρόταση υδρολογικού σχεδίου για τη λεκάνη απο... απορροής του ποταμού Εύρο, κάτι το οποίο υποτίθεται ότι παραβαίνει διάφορες ε, περιβαλλοντικές, περιβαλλοντικές οδηγίες, εγώ θέλω να εκφράσω τη διαφωνία μου. Δεν θα αναφερθώ ε, στο περιεχόμενο της απάντησης του Ισπανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο μελετά το θέμα και αξίζει τα μέλη της Επιτροπής να μελετήσουν την απάντηση του Ισπανικού Υπουργείου, διότι δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις στους αναφέροντες. Μιλούμε για ένα σχέδιο το οποίο είναι στην, ε, στα Σπάργανα, θα πρέπει να διατυπωθεί περαιτέρω, να τύχει περισσότερης επεξεργασίας. Αν το εξετάσουμε όμως αυτό το υδρολογικό σχέδιο, θα δούμε ότι προσπαθεί ε, να δώσει νέες γραμμές διαχείρισης επιδιώκοντας ισορροπία μεταξύ των διεκδικήσεων των διαφόρων επικρατιών και των διεκδικήσεων για το περιβάλλον και των διεκδικήσεων των χρηστών. Δεν είναι εύκολο να συγκεραστούν αυτά τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Όμως το Συμβούλιο για τα Ήδατα ε, ασχολήθηκε με το θέμα της λεκάνης απορροής του ποταμού που είναι και το ανώτατο όργανο που αποφασίζει ε, ε, ψήφισε 70 υπέρ 9 κατά 5 αποχές υπερψήφισε αυτό το υδρολογικό σχέδιο και το Συμβούλιο απαρτίζεται από εξέχοντα μέλη. Είναι μια έκθεση της 4ης Ιουλίου του 2013. Μέσα σε αυτές τις ευνοϊκές ψήφους, 72 ψήφισαν υπέρ, 8 από τις 9 αυτόνομες κοινότητες που εκπροσωπούνται έχουν υπερψηφίσει η Αραγωνία, η Ναβάρα, η Λαριόχα, η Καστήλη Λεόν, η χώρα των Βάσκων, η Κατάμπρια και η Κομμουνιδά Βαλενθιάνα. Μόνο η Καταλωνία καταψήφισε το υδρολογικό αυτό σχέδιο. Οκτώ από τις εννέα αυτόνομες κοινότητες το υπερψήφισαν και ήταν μια πολύ συμμετοχική διαδικασία για να καταλήξουμε σε αυτό. Αντίθετα με ό,τι λέει ο αναφέρον, 120 συνεδριάσεις με πάνω από 1.700 εκπροσώπους από διάφορες συλλογικότητες, ε, μήνες πολιτικής διαβούλευσης, δημόσιας διαβούλευσης, 6.000 συνεισφορές. Πάρα πολλά πράγματα έχουν συμπεριληφθεί στο έγγραφο. Είναι πολύ εξαιρετικά συμμετοχική η διαδικασία ε, βάσει της οποίας καταλήξαμε σε αυτό το υδρολογικό σχέδιο, το οποίο είναι απλά και μόνο ένα σχέδιο. Θα ε, τελειοποιηθεί έτσι περαιτέρω. Θέλω πολύ απλά να πω ότι εγώ είμαι από την Αραγωνία, όπου πολύ συχνά στα χωριά από τα οποία περνάει ο ποταμός Εύρο πρέπει να εφοδιάζονται τα χωριά από δεξαμενές και από βιτιοφόρα γιατί, γιατί δεν έχουν νερό ενώ το ποτάμι περνάει μέσα από το χωριό. Ε, δεν είναι δυνατόν. Έχουμε ε, σχέδια ε, βιολογικού καθαρισμού, επεξεργασίας λιμάτων, επαναχρησιμοποίησης ε, λιμάτων, αποκατάσταση των παρόχθιων περιοχών, ε, καταπολέμηση της ερήμασης, καταπολέμηση των ειδών που είναι εισβολής και βλάπτουν την τοπική χλωρίδα και πανίδα, κάτι το οποίο είναι όλο και πιο παρόν. Χρειαζόμαστε ε, περισσότερα ε, φράγματα γιατί μέρος της λεκάνης απορροής κάθε χρόνο πλημμυρίζει. Και τι γίνεται με τις οικολογικές κήτες, αυτό αυτά τα οποία λειτουργούν ως διάβλη, αν θέλετε, για το περιβάλλον. Η πρόταση αυτή ορίζει για πρώτη φορά τι σημαίνει οικολογική κήτη, οικολογικός διάβλος και ε, θεωρεί ότι είναι στρατηγική σημασία και μόλις εγκριθεί θα πρέπει όλοι να τη στηρούν και να τη σέβονται. Αυτός ο νομικός ορισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός από κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής πλευράς και η οικολογική διάβλη ε, προσδιορίζονται αυτά τα ελάχιστα ποσοστά για τους οικολογικούς διάβλους που θα πρέπει να προστατευτούν με πάση θυσία είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι σε άλλες περιοχές της Μεσογείου ή σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αυτές είναι πολύ σημαντικές βελτιώσεις και είναι αντικειμενικά αυτά τα στοιχεία. Εξού και δεν συμφωνούμε ε, με τους προλαλήσαντες και δεν πιστεύουμε σε καμία περίπτωση ότι αυτό το σχέδιο παραβαίνει την οδηγία πλαίσιο για τα νερά, ούτε για τους οικότοπους, ούτε για την περιβαλλοντική ευθύνη. Πιστεύουμε ότι αυτό το υδρολογικό σχέδιο πραγματικά είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας, θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση και όλες οι αυτόνομες κοινότητες εκτός από μία είναι αλληλέγγυες υπερασπιζόμενες το. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο ομιλητής. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες, οι οποίοι δυστυχώς για άλλη μια φορά πρέπει να έρθουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να εξηγήσουν κάτι το οποίο ε, είναι μέρος της κοινή λογικής και της δημοκρατικής διαδικασίας. Η διαχείριση των δημοσίων αγαθών βασίζεται στο δημόσιο συμφέρον και όχι στο ιδιωτικό συμφέρον. Και αυτή είναι η βασική παραδοχή που πρέπει να θέσουμε επιτάπητος. Πρώτον, δημοκρατικής πλευράς. Δεν μπορείτε να λέτε όταν, ότι έχει γίνει δημόσια διαβούλευση, όταν εδώ και πέντε χρόνια δεν έχει γίνει καμία τεχνική συζήτηση επί τούτου. Δεν μπορείτε να λέτε ότι, ότι εκπροσωπείτε συλλογικότητες, όταν οι συλλογικότητες που πλήττονται περισσότερο από αυτό το σχέδιο δεν τις ακούσατε, δεν τις καλέσατε, και δεν ε, εξετάσατε τις τοποθετήσεις τους που σας υποβάλλουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, από πλευράς συμμετοχικότητας και συμμετοχικής δημοκρατικής διαδικασίας το πρόβλημα είναι σοβαρό. Από πλευράς διαφάνειας το πρόβλημα είναι ακόμα σοβαρότερο και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανησυχήσει γι' αυτό. Διότι ιστορικά είναι μία από τις θεμελιώδεις συζητήσεις, τις βασικές συζητήσεις που κάνουμε στην Επιτροπή μας. Να άλλο ένα παράδειγμα γιατί χρειάζεται δημόσια, ανοιχτή, διαφανής συζήτηση και διαβούλευση. Τρίτον, αποσύρεται η συνάδελφος και δεν ακούει, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάτε για την αλληλεγγύη των αυτόνομων κοινοτήτων πότε θα ξεκινήσουμε να μιλούμε για την περιβαλλοντική ευθύνη και για την ευθύνη μεταξύ των γενεών. Πότε επιτέλους θα αρχίσουμε να ε, παίρνουμε στα σοβαρά τα χρέη που δημιουργούμε και που θα βαρύνουν τις μελλοντικές γενιές. Πότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα, αν είναι αναντίστρεπτες, θα τις πληρώσουν οι επόμενες γενιές και δεν θα μπορέσουν καν να μας ζητήσουν το λογαριασμό δεν μπορούμε να ξανά να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Στη διαχείριση του νερού έχουμε αρκετή εμπειρία και πρέπει να γνωρίζουμε πλέον ότι τέτοιου είδους πολιτικές δεν μπορούν να εφαρμόζονται πια. Έχουν τελειώσει. Σε 50 χρόνια το 80% των οικοσυστημάτων και ε, ε, ε, των, εδαφών στο Δέλτα θα έχει εξαφανιστεί αν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Τα νούμερα είναι πολύ απλά. Τρίτον, δεν μιλούμε για άλλο ένα υδρολογικό σχέδιο. Ξεκινά για άλλη μια φορά η συζήτηση επί της ουσίας. Η οποία πια είναι η συζήτηση επί της ουσίας. Η καινούρια κερδοσκοπική φούσκα που πάει να δημιουργηθεί. Είχαμε πρόσφατα την φούσκα με τα στεγαστικά και τα κατασκευαστικά στην Ισπανία και τώρα θα έχουμε κερδοσκοπική φούσκα γύρω από τα ύδατα γενικότερα και το νερό. Όλα αυτά αντιβαίνουν ε, στο δημόσιο συμφέρον, πλήττουν τις επόμενες τις μελλοντικές γενιές και Συμπερασματικά, ε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξή: Αυτό το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι η κοινή λογική. Η κοινή λογική όχι μόνο των Ισπανικών αρχών αλλά και των Ευρωπαϊκών αρχών. Εγώ συνεχίζω να έχω εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι και οι φίλοι από την πλατφόρμα από αυτή τη συλλογικότητα πιστεύουν στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιδείξει πολύ κοινή λογική ε, στα θέματα της διαχείρισης των υδάτων, πολύ περισσότερη και μεγαλύτερη από τις ε, εθνικές κυβερνήσεις. Ελπίζουμε η Επιτροπή να συνεχίσει να υπερασπίζεται το κοινό καλό, την κοινή λογική και το δημόσιο συμφέρον. Γιατί αυτά είναι το μήνυμο της λογικής. Ε, αν δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να καταδείξουμε τον επίγοντα χαρακτήρα των αιτημάτων μας, ε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν εγκριθεί αυτό το σχέδιο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκατασταθούν τα λάθη ε, που θα ε, προκληθούν από την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Ο κύριος Τρεμόσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα, δεν θα καταχραστώ το ότι μου δίνετε το λόγο. Θα μιλήσω μόνο δύο λεπτά. Καλωσορίζω την πλατφόρμα υπεράσπισης του Εύρω και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να έρθετε πολλές φορές ξανά στον οίκο μας. Πρώτον, θα πρέπει να αξιολογήσουμε το εξής. Η κείμενη νομοθεσία ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβλεπε το 2000, για το 2009 την έγκριση των υδρολογικών σχεδίων και των σχεδίων για τις λεκάνες απορροής των ποταμών. Όπως δυστυχώς συμβαίνει συχνά, δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση στην Ισπανία παρόλο που ε, δεχθήκαμε τις εγκλήσεις του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έλλειψη αυτή. Μιλούμε για αυτούς τους διάβλους που θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές αρδεύσεις. Εγώ μιλώ εξ ονόματος του φιλελεύθερου λαϊκού κόμματος της Καταλωνίας, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή και την κυβερνητική πλειοψηφία στην αυτόνομη κοινότητά μας. Θεωρούμε ότι το υδρολογικό σχέδιο περιορίζει σε λιγότερα από 3.000 ε, κυβικά εκατοστά το χρόνο, ώστε άνω των 11.000 κυβικών εκατοστών ε, να αφιερωθούν στην άρδευση στα ανώτερα ε, τμήματα του ποταμού, από εκεί που ξεκινάει δηλαδή. Αντί για λιγότερα από 3.000 κυβικά εκατοστά, εμάς θα μας χρειάζονταν 7.000 κυβικά εκατοστά και αυτό είναι μια επιστημονική άποψη και φαίνεται η διαφορά, η απόκληση. Από εκεί και πέρα η απάντηση που εδόθη δεν είναι η κατάλληλη και δεν δείχνει σωστή σχέση μεταξύ αρμοδίων διοικητικών αρχών, μεταξύ των διαφόρων αυτονόμων ε, κοιτοτήτων. Ε, εκφράζει μόνο την άποψη της πλειοψηφίας και η αυτόνομη κυβέρνηση της ε, Καταλωνίας ετέθη στο περιθώριο ενώ ήταν ισότιμος εταίρος στη λήψη των αποφάσεων. Εξού και εμείς απορρίψαμε συνολικά κάθε ένα αλλά και όλα μαζί τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας και έναν πολιτικό προβληματισμό. Με τον ε, ποταμό Τάγο, ο οποίος εκβάλλει στην Πορτογαλία, καμία ισπανική κυβέρνηση ποτέ δεν ε, είπε ότι θα ε, εκτρέψει το 70% των υδάτων για να το χρησιμοποιήσει το Ισπανικό κράτος ε, και τελικά θα φτάνει στο Δέλτα το Πορτογαλικό μόνο το 30% αυτό που θα έφτανε και που έφτανε νωρίτερα. Δεν είχε τολμήσει καμία Ισπανική κυβέρνηση να το κάνει αυτό σε μια ξένη χώρα την Πορτογαλία και δεν το έχει κάνει ποτέ. Ωστόσο αυτό κάνει στη δική μας περίπτωση. Έχουμε ανοίξει εκ νέου αυτό το θέμα του νερού θεωρώ ότι δίδονται κίνητρα λογικά και όλο και πιο έντονα υπέρ της πλήρης ανεξαρτητοποίησης του κράτους της Καταλωνίας. Αν ήμασταν ως Καταλωνία ανεξάρτητο κράτος θα μας σεβόταν περισσότερο η Ισπανική κυβέρνηση όπως σέβεται και την Πορτογαλία. Και ε, γι' αυτό καλό την Ισπανική κυβέρνηση και τις ε, περιφέρειες όπου κυβερνά το Λαϊκό Κόμμα να εξετάσουν αυτό το θέμα όχι όπως το εξέτασαν πριν από δέκα χρόνια. Ο Υπουργός τότε μιλούσε για στρατιωτικά βήματα προς την κοινότητα της Βαλένθια. Εμείς δεν είμαστε κατά της άρδευσης. Εγώ προέρχομαι από τη Λέριδα και γνωρίζω πόσο έχει ωφελήσει η άρδευση όλες αυτές τις κοινότητες εκεί. Όμως, τον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να ε, υποστηρίζουμε ότι μπορούμε ερημικές εκτάσεις να τις κάνουμε τόσο, ε, με τόση βλάστηση όσο να ήταν ε, στον Ατλαντικό με τις βροχοπτώσεις του θα πρέπει να εγγυηθούμε μία ελάχιστη κήτη στην εκβολή του ποταμού. Καλό το Ισπανικό κράτος να δει τα πράγματα υπό το φως των γνώσεων του 21ου αιώνα και ε, να αφουγκραστεί τα αιτήματα που αποτελούν την, τα αιτήματα που απηχούν την έντονη πλειοψηφία του καταλανικού λαού. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι γεωλόγος. Με τη δικτατορία του Φράγκο δεν κατάφερα να ασκήσω το επάγγελμα και άσκησα άλλο επάγγελμα. Εν πάση πτώση κάτι μου έχει μείνει από αυτά που σπούδασα στο πανεπιστήμιο τότε. Και πιο συγκεκριμένα έχω να πω το εξής. Έχω δει τόσες πολλές καταστροφές στη ζωή μου στην παράκτια ε, περιοχή ε, της Ισπανίας στη Μεσόγειο, όχι μόνο στην αυτόνομη κοινότητα της Καταλωνίας αλλά και αλλού πόσο κατέστρεψαν ε, το τοπίο. Και αυτό το οποίο έχω δει είναι ότι αυτοί που προκάλεσαν αυτές τις καταστροφές συμμορφωνόντουσαν με όλους τους νόμους, με όλες τις ε, οδηγίες και εκφωνούσαν ομιλίες άψογες, συμμετείχαν σε συζητήσεις με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Τελικά όμως έγινε χώρα, ε, έλαβε χώρα, σημειώθηκε αυτή η καταστροφή του φυσικού τοπίου στην παράκτεια ε, περιοχή της Ισπανίας. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επαγγελματίας για να το αντιληφθεί. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να σας εξηγήσουμε εδώ. Το δέλτα του ποταμού Εύρο ή Εύρος είναι ένα αγαθό που ωφελεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι κάτι το εξαιρετικά εύθραυστο και πρέπει να προστατευθεί. Πιστεύω ότι πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα όλης αυτής της ε, καταστροφής της παράκτιας περιοχής της Ισπανίας τις τελευταίες δεκαετίες και να μην αφήσουμε να μας εξαπατήσουν οι διάφορες ε, ρυθμίσεις, διατάξεις, ρήτρε νομοθετικές και μη ώστε να καταφέρουμε να σώσουμε το δέλτα του εύρου ε, τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Βεβαίως όταν καταστραφεί το ΔΕΛΤΑ ή όλα αυτά δεν θα είμαστε εμείς εκεί για να ε, μας ζητηθούν ευθύνε και να δώσουμε λογαριασμό. Ε, δεν θα ζούμε τότε. Εμείς ως σοσιαλιστές στηρίζουμε πλήρως την πλατφόρμα υπεράσπισης του, Δέλτα του Ποταμού Εύρου, τις πλατφόρμες κατά των φραγμάτων και των εκτροπών. Ε, θέλουμε να κινητοποιήσουμε όλους ενάντια σε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά απειλητικό και σε κάτι το οποίο βρίσκεται υπό πολύ έντονη απειλή. Εάν η δημοκρατία είχε την απαραίτητη δύναμη να τα βάλει ε, με το χρήμα και με την αγορά, θα ήταν απόλυτα βιώσιμη η λογική λύση. Δυστυχώς όμως τα χρόνια που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι βάρβαρα η κρίση κάνει την εξουσία του χρήματος να υπερισχύει έναντι της κοινή λαϊκής βούλησης την οποία εκφράζουν με δημοκρατικό τρόπο οι πολίτες. Εμείς ε, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ε, για το στρατόπεδο με το οποίο θα συνταχθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Κάρλος Ιτουργκάιθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ε, τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή Αναφορών. Δεν θα το επαναλάβω. Ευτυχώς την κοινή λογική την παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να τους ακούσουμε. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν άψογη, δεν μπορεί να αποφανθεί ε, μέχρι ότου ε, υποβληθεί το σχέδιο για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Εύρου και τότε θα αξιολογήσει κατά πόσο το σχέδιο αυτό συνάδει με την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως πρέπει να πούμε το εξής, να υπογραμμίσουμε ότι Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμειχθεί με τη διατύπωση αυτού του προσχεδίου, του υδρολογικού σχεδίου, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να καθυστερήσουμε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία και έτσι να υπάρξουν ακόμα περισσότερα ε, προβλήματα και λύσεις. Δεν σας άρεσε κύριε Ρομέρο όταν είπαμε ότι ε, πολλές αυτόνομες κοινότητες και η δικιά μου η Λαριόχα υπερψήφισαν αυτό το σχέδιο αλλά αντιμετωπίζουν και όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για την Καταλωνία αλλά και για τη χώρα των Βάσκων και για τη Λαριόχα και για την Αραγωνία. Προφανώς είναι πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν να νομίζετε ότι μόνο εσείς θα έχετε πρόβλημα και όχι εμείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πει πρέπει να ξέρει ότι οι αναφέροντες είχαν τα απαραίτητα ένδικα και νομικά μέσα στην διάθεσή τους για να ε, εκφραστούν και για να αναλάβουν δράση. Οι απαντήσεις του Υπουργείου είναι οι σωστές. Γνωρίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία είναι 29 Ιουλίου. Εάν προτρέξουμε ε, και απορρίψουμε κάτι το οποίο είναι στη φάση του προσχεδίου, ενώ το τελικό σχέδιο θα το έχουμε στις 29 Ιουλίου και τότε θα ξέρουμε αν πραγματικά υπάρχει παράβαση νομοθεσίας, νομίζω ότι θα προτρέξουμε ε, και επειδή θα βιαστούμε τελικά θα σκοντάψουμε. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι ε, ε, καλό είναι να επιτρέψουμε να ολοκληρωθούν οι διάφορες διαδικασίες χρονικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφανθούμε με ηρεμία για να δούμε ποια είναι τα βήματα τα συγκεκριμένα που κάνει αυτή τη στιγμή η, κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ η κυρία Έρανθ. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω τους αναφέροντες που, έρχονται, που έχουν έρθει μέχρι εδώ για να υποβάλουν την αναφορά αυτή. Εγώ έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Θαραγώθα. Ε, έχω σπουδάσει γεωγραφία και ε, έχω εξειδικευθεί στην ε, τοπογραφία. Μπορείτε να διαφωνείτε μαζί μου ή να συμφωνείτε, αλλά ε, πρέπει να γνωρίζετε ότι ξέρω επιστημονικά γιατί μιλάω και δεν μιλάω επειδή υπερασπίζομαι πολιτικά συμφέροντα και μόνο. Και μάλιστα είμαι και από το Λογρόνιο και όπως γνωρίζετε το σχέδιο αυτό μας αφορά και μας πλήττει άμεσα. Ξέρω το σχέδιο του Μπορέλ, λογικό σχέδιο είχε ονομαστεί τότε. Ήταν σχέδιο σοσιαλιστών και γι' αυτό ε, κατέληξε τα σκουπίδια. Μετά, αυτό όταν σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο, μετά είδα το υδρολογικό σχέδιο του Λαϊκού Κόμματο και τη κυβέρνηση Αθνάρ. Και μετά στα χρόνια του Θαπατέρο, των σοσιαλιστών και πάλι, δεν παρουσιάσε κανένα υδρολογικό ε, σχέδιο που να είναι σοβαρό. Ποτέ δεν παρουσίασε η κυβέρνηση Θαπατέρο ε, υδρολογικό σχέδιο που να είναι σοβαρό για μια χώρα η οποία ε, δεν έχει διαχειριστεί τα, ίδια τα, τα ενώ τα χρειάζεται τόσο πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι συμφωνεί με το σχέδιο λεκάνης απορροής του ποταμού ε, που παρουσιάζει η Ισπανία γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε και την Ευρωπαϊκή Οδηγία αλλά και την απόφαση του Δικαστηρίου του περασμένου Οκτωβρίου και πρέπει να διασφαλίσουμε έναν ε, οικολογικό διάβλο όπου θα προστατεύονται τα είδη ε, ώστε να συμμορφωθούμε με την νομοθεσία. Άκουσα πολλά πράγματα που με έχουν εκπλήξει σήμερα ότι δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της σκήτης του ποταμού κατά, τη διά, δια, δια τις διαφορετικές ε, περιόδους του χρόνου να έχουμε διαφορετικούς οικολογικούς διάβλους με διαφορετικές ποσότητες κυβικών εκατοστών νερού που θα πρέπει να διέρχονται αυτών. 800 κυβικά ε, ανά δευτερόλεπτο στο Δέλτα στις τελικές εκβολές τους καλοκαιρινούς μήνες και το φθινόπωρο και 150 κυβικά ανά δευτερόλεπτο στους μεγαλύτερους μήνες μέχρι το Μάρτιο. Δηλαδή, άρα ήδη το μελετήσατε το δέλτα του ευρώ, ενώ λέτε ότι δεν έχει μελετηθεί και ήδη από τη δεκαετία του 90. Και αυτό ισχύει όχι μόνο ε, στο δέλτα του Εύρου, στις εκβολές, αλλά και σε άλλα χωριά και σε άλλες περιοχές και στη δική μου κοινότητα, στην πόλη του Λογρόνια. Μην λέτε ότι δεν έχουν γίνει μελέτες, να πείτε ότι δεν σας αρέσουν οι μελέτες που ε, δεν έχουν γίνει, γιατί δεν ανταποκρίνεται αυτά που λέτε στην πραγματικότητα. Όταν θα έχουμε την έγκριση ενός σχεδίου, του υδρολογικού σχεδίου για τη λεκάνη απορροή στη Κουέγκα, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν το δούμε αυτό, τότε θα μπορέσουμε ε, να δούμε κατά πόσο θα εφαρμόσουμε διορθωτικά μέτρα και γι' αυτό λέγονται και διορθωτικά μέτρα γιατί ε, με αυτά δίνει μεγαλύτερη έμφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα που δεν ήταν δυνατόν να βγουν στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια την αρχική φάση της διαδικασίας. Να δουλέψουμε λογικά προτείνω και έτσι δουλεύουμε πάντοτε στη χωροταξία, στην τοπογραφία ε, και στη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Μας ασκείτε κριτική και λέτε ότι σε συνθήκες σκοταδισμού δουλεύουμε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Στην Ισπανία και στην Καταλωνία έχουμε νόμους εθνικούς της κεντρικής κυβέρνησης, περιφερειακούς της τοπικής κυβέρνησης, της αυτόνομης, της αυτόνομης κοινότητας και ε, ε, αυτοί οι νόμοι λένε ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Μην μου λέτε ότι δεν έχουμε τέτοιους νόμους και διατάξεις. Είναι σαν να λέτε ότι πήρατε κλίση και πρόστιμο επειδή κάνατε οδική παράβαση και ότι δεν είναι σωστό. Σε κανέναν δεν αρέσει να παίρνει κλίση, να του κόβει κλίση ο αστιφύλακα, αλλά πρέπει να την πληρώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Μη λέτε πράγματα που δεν, αντιστοιχούν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και μάλιστα αυτό που με ενοχλεί είναι που ιδιοποιείστε το ποτάμι αυτό. Φαίνεται σαν να ανήκει σε κάποιον συγκεκριμένα. Δεν ισχύει αυτό. Κανείς ε, δεν έχει αποκλειστικό δικαίωμα στο ποτάμι αυτό. Ο Εύρος πηγάζει από την Καντάβρια και εκβάλλει στην Ταραγώνα. Όλες ε, οι επικράτειες, όλα τα εδάφια, όλες οι αυτόνομες κοινότητες έχουν ίσα δικαιώματα και πρέπει να ε, πούν την ε, άποψή τους. Εσάς δεν σας αρέσει και έχετε παρεμποδίσει ε, την εφαρμογή αυτού του σχεδίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ερμηνεύετε με συμβιλικό τρόπο την άρδευση και κάνετε την ύπουλη ερώτηση του ποιος πληρώνει τις αρδεύσεις. Τις αρδεύσεις τις πληρώνουν όσοι αρδεύουν. Υπάρχει νόμος που τα ρυθμίζει όλα αυτά και πληρώνουν τις αρδεύσεις και όσοι αρδεύουν στο Δέλτα του Εύρου, εσείς δηλαδή που έχετε ε, οποροκυπευτικά ε, και διάφορες καλλιέργειες στο Δέλτα του Εύρου και εσείς χρησιμοποιείτε το ποτάμι για τη γεωργία. Μην λέτε ότι το κάνουν μόνο οι άλλοι. Η χώρα μας είναι παραγωγός οποροκυπευτικών και πρέπει να έχει το δικαίωμα να ποτίσει σε όλα τις αρδεύσιμες εκτάσεις. Στην Ισπανία οι τεχνικές άρδευσης νερού είναι οι πιο εξελιγμένες, οι λιγότερο σπάταλες, οι πιο ε, προχωρημένες επιστημονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να επιβληθεί από την Κομισιόν μείωση κατά 25% της άρδευσης στην χώρα μας όπως απαιτείται γενικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εμείς ήδη ως χώρα έχουμε καταφέρει αυτή την εξοικονόμηση κατά 25% εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, σεβόμαστε ε, την οδηγία για τα πτηνά και για την περιβαλλοντική ευθύνη. Δεν είναι περιβαλλοντικό το πρόβλημα, είναι πολιτικό. Αυτό το οποίο σας ενοχλεί είναι ε, η απόφαση του κόμματος της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κυρία Χάουγεν. Θα είμαι πολύ σύντομη να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που έκαναν εξαιρετική παρουσίαση με κάπως ηλικιωμένη και ήδη στο σχολείο είχα μάθει για τον Έμπρο και για αυτή την περιοχή που είναι τις ωραιότερες της Ευρώπης και είναι καλό που έχουμε και υπερασπιστές της περιοχής ε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτός από τους αναφέροντες για τις ε, σαφείς απαντήσεις. Είναι σαφές ότι πολλά είναι τα συμφέροντα που πάνε να αποδυναμώσουν την ενωσιακή νομοθεσία, ε, να την αποδυναμώσουν. Ε, Παρ' όλα αυτά Έχουμε σαφή ε, απάντηση της Κομισιόν, έχουμε ξεκάθαρη νομοθεσία, πρέπει να την υπερασπιστούμε και να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ε, μείνουμε στις ε, συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες και τους νόμους. Ευχαριστούμε πάντοτε χαιρόμαστε για την ξεκάθαρη γλώσσα που ακούσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Μιράντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τους αναφέροντες και τις αναφέρουσες, οι οποίοι μπόρεσαν να έρθουν σε αυτή την Επιτροπή που αφογκράζεται τις ανάγκες των πολιτών. Έχουν ξαναέρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μοιραστούν μαζί μας αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει τις απαρχές του ε, σε κάπου πολύ μακριά. Η διαχείριση των υδάτων στην Ισπανία δεν είναι μοντέλο για την Ευρώπη. Το 1999 όταν χτίστηκε το φράγμα της Ούμια, το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είχε κάνει αντιγραφή και επικόλυση της μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου που είχε γίνει σε μια επαρχία της Ανδαλουσίας, ε, όσα, και το είχαν κάνει αντιγραφή μόνο όσα υποτίθεται μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου για άλλη αρχή στη Γαλλικία που είναι βόρειο-δυτικά και δεν έχει καμία σχέση το κλίμα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα ερμηνεία νομοθεσία, είναι θέμα εφαρμογή αυτή. Δεν είναι μόνο πολιτικό το ζήτημα, είναι και οικονομικό. Διακυβεύονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα, τα οποία είναι άρρηκτα δεμένα με το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο έχει την πλειοψηφία, και έρχονται στην Επιτροπή μας ε, αυτοί του Λαϊκού Κόμματος μόνο για να υπερασπιστούν την κυβέρνησή τους. Μόνο όταν ε, ε, υπάρχει θέμα που τους απασχολεί προκειμένου να προστατεύσουν τα ε, συμφέροντα τα οποία υπερασπίζονται ούτως ή άλλως και έρχονται εδώ, ε, ανοίγουν το μικρόφωνο, λένε αυτό που έχουν να πούν και φεύγουν και δεν ακούνε καν τον αντίλογό μας ούτε μένουν για να δευτερολογήσουν και δείχνουν την έλλειψη σεβασμού εναντί αυτής της Επιτροπής. Εγώ εκπροσωπώ δύο κόμματα, την Δημοκρατική αριστερά της Καταλωνίας αλλά και την ε, διοικητική ε, μεταρρύθμιση της Αραγωνίας. Ε, έχουμε μεγάλη συνένεση και έχουμε πλήρη ομόνια απόψεων. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αξιολόγηση. Υπάρχει έλλειψη συμμετοχής, έλλειψη επιστημονικών στοιχείων, μονομερή σύνταξη εκθέσεων και δεν ε, ελήφθη υπόψη η άποψη των 100.000 κατοίκων. Συμφωνώ με την προλαλή σας, το ποτάμι και τα ποτάμια δεν ανήκουν σε κανέναν. Ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει ε, να έχουμε αυστηρότητα στην προσέγγιση μας. Υπάρχει και προηγούμενο η διαδικασία επί παραβάση που παραμένει ανοιχτή ε, στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθήσει πολύ στενά το ζήτημα αυτό, γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον ολόκληρης της χώρας και αυτό που διακυβεύεται επίσης είναι ε, η αξιοπιστία των ίδιων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιγγελάνχελ Μαρτίνεθ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, για να είμαι ειλικρινής, μετά από την ε, παρέμβαση ε, του συναδέλφου Όλιος, δεν θα χρειαζόταν να πω τίποτα άλλο. Να πω μόνο ότι συμφωνώ 100% με τον προηγούμενο ομιλητή. Όμως, επειδή και άλλοι πήραν το λόγο και είπαν άλλα πράγματα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ακουστεί. Είμαι από τη Λαμάντσα και γνωρίζω τα του νερού. Είναι ένα από τα πιο εφιαλτικά προβλήματα που μπορεί κάποιος να, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του νερού. Υπάρχουν νόμιμα συμφέροντα, θεμητά συμφέροντα που κάνουν τη μία αυτόνομη κοινότητα να επιτίθεται στην άλλη και αντιστρόφως. Εάν θέλουμε να έχουμε αλληλεγγύη και δυναμισμό, ε, πρέπει να το προσπαθούμε πάρα πολύ, διότι έχουμε δυσκολευθεί πολύ στο παρελθόν να επιβάλλουμε αυτή την αλληλεγγύη και αυτό το δυναμισμό, αποφεύγοντας το λαϊκισμό, αλλά και τους εκβιασμούς, τους εκβιασμούς ενίοτε που έχουν υπάρξει και γνωρίζετε τα παραδείγματα του παρελθόντος ε, των εκβιασμών μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, ε, των αυτόνομων κοινοτήτων ή και των ε, πολιτικών παρατάξεων. Αδιαφυσβήτητα όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ποια θα είναι, πώς μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση ενός ποταμού για όλους. Και φυσικά μέσα στην αξιοποίηση ε, του ποταμού τίθεται ε, και το περιβαλλοντικό ζήτημα, η περιβαλλοντική προστασία, η οποία μπορεί μάλιστα και να επικρατεί έναντι άλλων ε, εκμεταλλεύσεων. Εγώ είμαι από τη Λαμάντσα και έχω ασχοληθεί ιδιαίτερως με το θέμα του ποταμού Τάχο ή Τάγο ο οποίος εκβάλλει στην Πορτογαλία και αναφέρθηκε νωρίτερα. Δεν είναι δυνατόν ένα ποτάμι να διασχίζει εδάφη και σε αυτά τα εδάφη να πεθαίνει ο κόσμος από τη δίψα και να προβάλλεται το επιχείρημα ότι ε, πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο το ποτάμι για να μην χαλάσει το δέλτα του. Εκεί που τελειώνει μετά από ε, τόσο μεγάλη απόσταση. Και αυτή ήταν η κατάσταση στη Λαμάντσα. Επί ολόκληρες ε, στη Λαμάντσα, στα χωριά έβλεπε ο κόσμος τον, ε, το ποτάμι να περνάει από μπροστά του και δεν μπορούσε να αρδεύσει και πεθαίναμε από τη δίψα γιατί εκβάλλει ε, στην Πορτογαλία και πρέπει το Δέλτα να παραμείνει ως έχει και πρέπει το ποτάμι να μην, να μην το αγγίξει κανείς. Ε, δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. σε κοινοτικό επίπεδο καταφέραμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια σειρά κανόνων που να είναι δεσμευτικοί για όλους, που να υποχρεώνουν όλους. Συμφωνώ με αυτά που λέει η κυρία Μιράντα. και συμφωνώ ότι δεν είναι δυνατόν οι του Λαϊκού Κόμματο να έρχονται εδώ, να λένε το παραμύθι του, να φεύγουν και να μην ακούνε ε, τι έχουμε να πούμε εμεί και να μην δευτερολογούν και να μην ακούν τη δική μα δευτερολογία. Είναι πράγματι έλλειψη σεβασμού αυτού. Σε κάθε περίπτωση, το υδρολογικό ε, σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και το οποίο υπερασπίστηκε η κυρία που καθόταν απέναντί μου, ε, κατέληξε στον κάλαθο των αχρήστων ε, γιατί δεν πληρούσε τίποτα από τα δέοντα. Αυτό δεν είναι ένα προηγούμενο που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας. Δεν δόθηκε προτεραιότητα στην τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση εμείς συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της πλατφόρμας υπεράσπισης του ΔΕΛΤΑ. Δεν συμφωνούμε με αυτούς που λένε ότι δεν υπήρξε συμμετοχική διαδικασία. Είναι σαν να μας λένε ότι οι φωτογραφίες με τους χιλιάδες διαδηλωτές είναι ψέματα. Τους έβγαλαν στον δρόμο να διαδηλώσουν και δεν ήξεραν οι άνθρωποι, δεν είχαν ενημερωθεί γιατί διαδήλωσαν. Αυτό σημαίνει κινητοποίηση, συμμετοχή, διαδήλωση, ενημέρωση, επικοινωνία. Ορίστε η φωτογραφία. Βλέπετε πόσο κόσμο είναι εκεί και διαδηλώνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμμετοχή ενώ έχει πλημμυρίσει ο δρόμος. Τι είναι, είναι πλαστογράφηση τη φωτογραφία, έχετε έχουμε κάνει κολάζ, υποτίθεται πώς λέτε ότι δεν έχει συμμετάσχει η κοινή γνώμη στη διαμόρφωση όλων αυτών. Ναι, έχει υπάρξει επικοινωνία, έχει υπάρξει ενημέρωση. Επιτέλους, να πούμε την αλήθεια. Η πλατφόρμα υπεράσπισης είναι εδώ γιατί ακριβώς εκπροσωπεί την λαϊκή κινητοποίηση. Όσο δεν συμφωνώ με το Λαϊκό Κόμμα, τόσο δεν συμφωνώ και με εσά που λέτε ότι δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμο. Όχι, έχει υπάρξει ενημέρωση, έχει υπάρξει επικοινωνία, έχει υπάρξει κινητοποίηση. Α ελπίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, τηρήσει τις υποχρεώσεις της και εμείς θα στηρίξουμε ε, την προστασία του περιβάλλοντος. Όμως το ποτάμι δεν ανήκει μόνο στο δέλτα του και σε όσους έχουν το δέλτα του και τις εκβολές του και οι άλλοι έχουν δικαιώματα όσοι είμαστε στο, κατά τη διαδρομή του ποταμού. Δεν μπορεί να λυθεί όλο αυτό το πρόβλημα με ένα μόνο τεχνικό και σύγχρονο τρόπο, ούτω ώστε να είναι όλοι απολύτως ικανοποιημένοι. Τι θέλετε δηλαδή, για να μην θέλετε να μας διώξετε από εκεί που μένουμε, οι επικράτειές μας και οι περιοχές μας πεθαίνουν από τη δίψα. Και δεν γίνεται να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό από ένα πετάμι που περνάει από τη γη μας. Θέλετε να εγκαταλείψουμε τη γη μας και να έρθουμε να κάτσουμε στο κεφάλι σας ε, ε, εκεί σε εσά τις εκβολές του ποταμού. Γιατί αυτό θα αναγκαστούμε τελικά να κάνουμε λόγω της τεράστιας ξηρασίας όταν δεν μας αφήνεται καθόλου να αρδεύσουμε. Εν πάση περιπτώσει κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι πρέπει να βρούμε ένα σωστό σημείο ισορροπίας για να μπορέσουν όλοι να χρησιμοποιήσουν το νερό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσανώνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έφτασα καθυστερημένος γιατί είχα κάποιες συνειλημμένες υποχρεώσεις, δεν κατάφερα να ακούσω την παρουσίαση. Άκουσα όμως τα προβλήματα για τα οποία, στα οποία εφερθήκα εδώ στον φορά το ποταμό Έμπρο. Άκουσα πολλές φορές ε, τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χρήση των υδάτων ε, των ποταμών. Εγώ προέρχομαι από μία επαρχία στην ε, βόρειο-ανατολική Ιταλία όπου έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα. Χθες μάλιστα υπέβαλα ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ασχοληθούμε περισσότερο με τη χρησιμοποίηση των υδάτων από την επαρχία του Μπελούνο, βόρεια από τη Βενετία, περιοχή στην οποία προβλέπονται 100 υδροελεκτρικοί σταθμοί. Και καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία πραγματικά χρησιμοποιείται και πρώτα θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Μάλιστα χάρη σε κάποια κίνητρα που έχουν δοθεί για να νεώσουμε πηγές ενέργειας, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ επιχειρήσει οι οποίε θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή αυτή χωρί να γνωρίζουμε όμω ακριβώ ποιε θα είναι οι περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με ένα μεγάλο άλλο ποταμό στην Ιταλία, τον Ιταλό Πιάβε, τον ποταμό με συγχωρείτε Πιάβε. Στην περιοχή αυτή αντιμετωπίζουμε ξηρασία εδώ και ένα χρόνο. Από το Σεπτέμβριο του 2011 και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012 είχαμε κάποιες ε, κάποια πάρα πολύ έντονα, έντονες επιπτώσεις ε, ξηρασίας. Υπήρξε μια ιδιαίτερη χρησιμοποίηση των υδάτων του ποταμού αυτού και υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ε, διαδήλωσαν, οι οποίοι εκφράστηκαν κατά της χρησιμοποίησης των υδάτων του ποταμού αυτού. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε όχι μόνο τον ποταμό αυτό, αλλά και όλη τη γύρω περιοχή προστατεύεται από την Natura 2000 και δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε στους πολίτες τα ελάχιστα είδετα από το ποταμό αυτό για ζητήματα άρδρευσης. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αξιολογήσουμε πάρα πολύ καλά την κατάσταση προτού γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αν οι παρεμβάσει αυτέ πραγματικά θα οδηγήσουν σε ωφέλη όσον αφορά τι τοπικέ κοινότητε, γιατί Μπορεί ενδεχομένως βραχυπρόθεσμα να έχουμε όντω κάποια ωφέλη, να δούμε κάποιες βελτιώσεις, αλλά πολύ φοβάμαι ότι μακροπρόθεσμα στη συνέχεια ενδεχομένως να καταλήξουμε σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε επιζήμιες συνέπειες όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την τοπική οικονομία. Κάθε φορά λοιπόν που προχωρούμε σε τέτοια έργα ή σαν αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν στην Ιταλία, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουμε έπειτα στην πρώτερη κατάσταση. Είναι, πρόκειται για μία αναστρέψιμα έργα ουσιαστικά. Η έκκληση λοιπόν που κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και προς όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά είναι η ακόλουθη. Ας μην προχωρούμε πάρα πολύ γρήγορα, ας μην προχωρούμε βιαστικά. Υπάρχουν ε, πολλές περιπτώσεις, έκδηλες περιπτώσεις στην Ευρώπη που έχουν αντιμετωπιστεί πάρα, πάρα πολλά προβλήματα ακριβώς επειδή κάποια έργα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, πολύ βιαστικά χωρίς να έχουν γίνει απαραίτητες περιβαλλοντικές ε, μελέτες, χωρίς να έχουμε αφουγκραστεί πρώτα τους, τοπικέ ε, τις τοπικές κοινότητες, χωρίς να γίνει δηλαδή μια δημόσια διαβούλευση. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι θα πρέπει στο μέλλον τουλάχιστον να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξολογήσεις και να καταφέρουμε να ατενίσουμε καλύτερα το μέλλον, να δούμε ποιες θα είναι οι μελλοντικέ περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πολλά πράγματα τα οποία βραχυπρόθεσμα οικονομικά εμφανίζονται θετικά, στο μέλλον μακροπρόθεσμα μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματικές καταστροφές όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την τοπική κοινότητα και την τοπική οικονομία. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους αναφέροντες για το τελικό γύρο παρεμβάσεων που θα είναι σύντομος, θέλω να διευκρινίσω το εξής ως προς την κυρία Έρανθ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είπε ότι στηρίζει το υδρολογικό σχέδιο. Είπε ότι περιμένει την έγκριση του σχεδίου από πλευράς Ισπανικών αρχών και τότε θα αποφανθεί αν συμφωνεί ή όχι αλλά επιτρέψαμε να έρθουν οι αναφέροντες για να έχουν περισσότερες λεπτομερίες και περισσότερες πληροφορίες. Έχετε εσείς το λόγο εν συντομία για να μπορέσουμε να εξάγουμε τα βασικά συμπεράσματα και να προχωρήσουμε. Εκτός μικροφώνου, κύριος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που έγινε η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε ε, ε, εσάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθατε. Ευχαριστούμε τα μέλη της Επιτροπής. Ε, αναφορών. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε σύγκρουση. Θέλουμε απλά να σημάνουμε το καμπανάκι του συναγερμού πριν είναι πολύ αργά. Από το 2000 το δουλεύουμε αυτό και το λαϊκό κίνημα υπάρχει από το 1963, διότι ο δικτάτορας ήθελε πρώτα να εκτρέψει ε, το ποτάμι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, καθημερινοί άνθρωποι, δεν είμαστε ακραίοι. Έχουμε μία συνταξιούχο και είμαστε τέσσερις που δουλεύουμε, είμαστε εργαζόμενοι, πήραμε άδεια προσωπική διακοπών για να έρθουμε και αύριο θα ξαναπάμε στα γραφεία μας να δουλέψουμε. Εάν πρέπει να υποφέρουμε, θα υποφέρουμε, γιατί ζούμε στο Δέλτο και ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε, εμείς σε όλες τις συνεδριάσεις ε, της ε, Συνομοσπονδίας ε, εξέτασης ε, του θέματος του ποταμού Εύρου εμείς ήμασταν παρόντες και αυτή την κυρία δεν την έχουμε δει ποτέ. Φαίνεται ότι είναι συνήθειό της να έρχεται να βγάζει ένα λόγο και μετά να φεύγει. Δεν μπορεί να γίνει αντιπαράθεση απόψεων. Δεν μπορούμε να πούμε έχει κάνει λάθος όταν κάποιος λέει κάτι και μεταφέρει και δεν ακούει. Υπάρχει μια μελέτη του 2007 που μπορεί να είναι αμφισβητήσιμη, που μπορεί να, να τροποποιηθεί, να πρέπει να τροποποιηθεί, αλλά δεν συζητήθηκε ποτέ, το μπήκε στο περιθώριο. Εάν δεν βελτιωθεί η, η κήτη και ο διάβλος, ο οικολογικός, το μέλλον του Δέλτα είναι ανύπαρκτο και αυτό είναι ευθύνη και της Ισπανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μην κλείσετε το θέμα. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να το συνεχίσετε, αλλά μην μας το κλείσετε. Σας παρακαλούμε. Ε, κάνετε ό,τι μπορείτε, θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά να παραμείνει το θέμα ανοιχτό. Μία κυβέρνηση μπορεί να σχεδιάσει με αποτελεσματικό τρόπο ή να ε, μη σχεδιάσει με αποτελεσματικό τρόπο δεν είναι μια απόλυτη καταστροφή. Κανείς δεν πεθαίνει αυτή τη στιγμή για κανένα λόγο. Να γίνει σωστή εφαρμογή το, της νομοθεσίας από το Ισπανικό κράτος και την Ισπανική κυβέρνηση. Αυτό ζητούμε. Ο Πρόεδρος. Θα κάνω ένα προσωπικό σχόλιο. Έχουμε καθυστερήσει. Αυτό δεν είναι σπάνιο. Συμβαίνει συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, έχουμε καθυστερήσει, έπρεπε να είχαμε εγκρίνει τα υδρολογικά σχέδια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και η επόμενη αναφορά έχει να κάνει με τον ποταμό ε, Τάγο. Γιατί καθυστέρησαν, γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν μπει στην κερδοσκοπική φούσκα των στεγαστικών δανείων και των, ε, της οικοδομής και των κατασκευών. Δεν ήταν στην ατζέντα τα θέματα του νερού. Γι' αυτό παρενέβησαν τελικά τα δικαστήρια. Έχουμε τώρα αυτή την ευκαιρία και χαίρομαι διότι αυτή η αναφορά θα μας επιτρέψει να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί το υδρολογικό αυτό σχέδιο, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να συνάδει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αυτό είναι και το πιο θετικό που θα μπορούσαμε να πετύχουμε άλλωστε. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων βασίζεται στις αρχές της εξοικονόμησης, της διαφάνειας, της λαϊκής συμμετοχής, ε, του σεβασμού στο περιβάλλον ε, και λοιπά Όλη, όλος ο διάβλος, όλη η κήτη θα διαμορφωθεί και θα χαρακτηριστεί με βάση αυτές τις παραδοχές. Ζητώ λοιπόν από τους συντονιστές, από όσους έχουν υποφορτιστεί με αυτό το ε, καθήκον, να μελετήσουν αυτή τη δυνατότητα προστασίας του δέλτα του ποταμού Εύρου, το οποίο είναι ένα από τα πιο πολύτιμα οικοσυστήματα της Μεσογείου. Ξέρετε, οριζόνες έχουμε στα δέλτα των ποταμών πάντοτε και είναι πασίγνωστο το ρύζι που παράγεται εκεί εδώ και χιλιετίες. Είναι μια περιοχή εξαιρετικά πολύτιμη από όλες τις απόψεις και σε όλα τα επίπεδα. Ελπίζω ότι όλοι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πράγματι προτείνει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, ώστε ε, να δουλέψουμε όλοι για να δούμε ότι πράγματι το σχέδιο συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Άπαξ και παρουσιαστεί και όταν παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο και όχι το προσχέδιο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πράγματι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίζει να εξετάζει το θέμα. Εάν δεν έχετε άλλα σχόλια, κλείνουμε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και πάμε σε άλλη λεκάνη απορροής, τη λεκάνη απορροής του ποταμού Τάχο. Eh. Περνάμε στην αφορά 834-2012 του Μιγγέλ Άγχελ Σάντσες Πέρε. Ο κύριος Δανιέλ Μαρτίνες θα μας κάνει μια παρουσίαση της αναφοράς αυτής εξ ονόματος του αναφέροντος και όλων όσων υπέγραψαν την αναφορά αυτή. Δίνω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο των τον για πέντε λεπτά. Ε, Καλημέρα σας. Θα θέλω καταρχάς να διευκρινίσω ότι πρόκειται για μια κοινή αναφορά. Θα πάρει κι άλλο το λόγο. Είμαι ο Ντανιέλ Μαρτίνεθ, αναφέρον από την Ενωμένη Αριστερά. Σας ευχαριστώ καταρχάς που με δέχεστε και χαιρόμαστε διότι η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ποταμός Τάγο. Θέλουμε η Επιτροπή να επιτηρήσει στενά την διαμόρφωση και διατύπωση του υδρολογικού σχεδίου ώστε να τηρούνται αυστηρά οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι για να αντιμετωπίσει την ολιγορία των Ισπανικών αρχών, ώστε ο ποταμός Τάγος να σταματήσει πλέον να είναι ε, μία ε, χωματερή. Καλημέρα σας. Και εγώ έρχομαι από τις παρόχθιες περιοχές του ποταμού Τάγο, η Τάχο, ένας το μεγαλύτερο ποτάμι της ε, ε, Ισπανίας, το οποίο πηγάζει από τα Ισπανικά βουνά και εκβάλλει στον Ατλαντικό ωκεανό στην Πορτογαλία. Ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε την βοήθειά σας. Τέσσερις δεκαετίες χείρις της διαχείρισης από τις διάφορες ισπανικές κυβερνήσεις μας οδήγησαν τελικά να μην έχουμε καν ποτάμι. Έχουμε ένα ποτάμι που είναι θνίσκον, ε, χωρίς νερά να κυκλοφορούν, χωρίς κήτη ε, ε, που να ρέει τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Και μάλιστα θέλει η Ισπανική κυβέρνηση να κάνει εκτροπή και φράγμα και να πάνε σε άλλη λεκάνη υδρολογική τα ελάχιστα νερά που έχουν μείνει. Θα το χάσουμε το ποτάμι. Και τι θα χάσουμε τελικά. Ε, δεν θα χάσουμε μόνο τα νερά, την ενέργεια, αλλά και ένα στοιχείο πολιτισμού της επικράτησας. Ένα ε, σάξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται διάφοροι υδροβιότοποι, δάση, ε, παραποτάμια βλάστηση. Το ποτάμι είναι ζωή, είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιστορίας μας, αλλά πρέπει να αποτελεί και μέρος του μέλλοντός μας. Εδώ και 45 χρόνια η Ισπανία αποφάσισε να εκτρέψει το 80% της βασικής κήτης του ποταμού Τάχο προς άλλη λεκάνη απορροής που θα εκβάλει τελικά στην Μεσόγειο. Και, χρόνια, ε, και κάποια χρόνια, όπως την περασμένη χρονιά, αποφάσισε να εκτρέψει το 100%. Εκεί χύνονται τα λίματα της Μαδρίτης και άλλων. Ε, χύνονται λίματα άνω των 6,5 εκατομμυρίων ε, κατοικών. Και τελικά με όλη αυτή τη δράση αυτά τα καθερά ναρά έχουν μετατραπεί σε μία μαύρη κοιλίδα. Εκεί όπου πηγάζει ο ποταμός, ε, τα νερά αυτά πηγαίνουν στις αρδεύσεις ε, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών οι οποίες φαίνονται πολύ όμορφες και τελικά σε εμάς καταλήγουν ως νερά τα λίματα της ε, Μαδρίτης περνάει και από το Τολέδο, η Κίτη φτάνει στα ελάχιστα επίπεδά της στην Αραχουέθε και τελικά περνάει από τα Ταλαβέρα Ντελαρέινα. Όλες αυτές οι περιοχές και πόλεις που σας αναφέρω είναι πόλεις απαράμιλου κάλους και έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία κληρονομιάς από την UNESCO. Πρέπει, σας δείχνουμε φωτογραφίες για να καταλάβετε πώς ήταν και πώς είναι ο, τάγος, ο τάχο, ο ποταμός αυτός. Η κατάστασή του δεν είναι αυτή που περιγράφεται στα επίσημα έγγραφα της επίσημης ισπανικής κυβέρνησης. Ε, σας καλούμε να λύσετε το σχέδιο και να λάβετε μέτρα. Στο προσχέδιο της δημόσιας διαβούλευσης έχουμε έγγραφα, έχουμε μελέτες, έχουμε έρευνες που υποστηρίζουν την άποψή μας. Για το ποτάμι αυτό η Ισπανική κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να αξιοποιεί στο έπακρον τις εξαιρέσεις μόνο και τις παρεκκλήσεις της οδηγίας για να πετύχει αυτό που θέλει. Και παρόλο που δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί αυτό το νερό, υποτίθεται ότι θα δαπανήσει η Ισπανική κυβέρνηση 5 δις ε, για το έργο αυτό. και υποτίθεται ότι θα έχουμε 2,4 ε, δις ευρώ για την αφαλάτωση. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Και θα έχουμε ανταλλαγή δικαιώματος χρήσης του νερού. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά ύποπτα. Τι θα γίνει με το ποτάμι. Θα έχουμε αυτά τα 2,4 δις για αφαλάτωση χωρίς να χρησιμοποιούνται ε, τα της ακτής. Παραβαίνει η Ισπανική κυβέρνηση και την, οδηγία, την πλαίσιο και στο πνεύμα και στο γράμμα της. Περνάει από ε, τρία σημεία, τα Λαδέρα Ντελαρέινα, το Λέδο και Αραγχουέθ, σε αυτά τα τρία σημεία δεν θα υπάρχει οικολογική κήτη, γιατί η Ισπανική κυβέρνηση για αυτά τα, για αυτά τα σημεία το ονομάζει νομική κήτη, δηλαδή η ελάχιστη δυνατή ή ανύπαρκτη. Θέλει ε, το πλεόνασμα το υδάτινο να υπάρχει κυρίως εκεί όπου πηγάζει ο ποταμός για να μπορεί να το διοχετεύει στην άρδευση. Αυτό επιθυμεί η Ισπανική κυβέρνηση. Η Επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει να περιμένουμε μέχρι το 2015 όπου θα εγκριθεί τελικά Τελικά υπάρχει ο κίνδυνος για άλλη μια χρονιά ο ποταμός αυτός να παραμείνει στο περιθώριο, η Ισπανική κυβέρνηση να κερδίζει συνεχώς χρονικές αναβολές και μεταθέσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νύπτει τα σχήρας της. Θα πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι βάσει το στοιχείο της δεν είναι ξεκάθαρο πώς τα πτηνά και οι υδροβιότοποι πλήττονται ξεκάθαρα από το σύστημα διαχείρισης των ποταμών. Κοιτάξτε, όταν έχουμε υδροβιοτόπους ε, που συνδέονται με τα ποτάμια και το ποτάμι δεν έχει νερό ή αν έχει ελάχιστο νερό και χείριστης ποιότητας ε, μολυσμένο, ε, πώς είναι το να υποστηρίζετε ότι δεν πλήττονται τα πιτινάκια και οι υδροβιότοποι. Νομίζω ότι είναι προφανής ο συσχετισμός. Κοιτάξτε, 166 ε, σημεία εξετάστηκαν μόνο από τα χιλιάδες που θα έπρεπε να εξεταστούν. Είναι σαν να μην γνωρίζουν γιατί μιλούν. Και αν δεν αρκούν όλα αυτά, τις επόμενες εβδομάδες θα υποβάλουμε αποδεκτικά στοιχεία και εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έγγραφο που έθεσε προς δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση της Ισπανίας αναγνωρίζει ότι πολλαπλά κομμάτια του ποταμού Τάγου δεν θα ανακτήσουν την προτέρα επαρκή τους κατάσταση ούτε καν από το 2026 και μετά. Άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος του υδάτινου όγκου αποθηκεύεται για να εκτραπεί προς άλλη λεκάνη απορροής. Μπορεί το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν να κοιτούν από την άλλη μεριά και να στρέφουν τα νότα τους προς αυτή την τραγική κατάσταση ε, που έχει δημιουργήσει η Ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να εποπτεύσετε στενά την Ισπανική κυβέρνηση, θέλουμε να παρακολουθήσετε στενά κατά πόσο εφαρμόζεται βήμα προς τη βήμα η Ευρωπαϊκή Οδηγία, όλες οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικές με το θέμα ε, στην Ισπανία τον ποταμό Τάχο τον έχουν καταδικάσει. Ελπίζουμε να μην τον καταδικάσετε και εσείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ ο κύριος Βαλέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και τις ανησυχίες σας, όπως είπα και στην προηγούμενη αναφορά, Τώρα το βασικό είναι ότι έχουμε σχέδιο ε, προκαταρκτικό που θα σχολιαστεί. Και όπως προβλέπει η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, θα ενημερωθεί η Ισπανική κυβέρνηση σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το πρώτο σχέδιο. Η οδηγία πλαίσιο επίσης προβλέπει ότι θα ε, αξιολογήσουμε τα έτοιμα σχέδια που έχουν υποβληθεί στην Κομισιόν. Ένας Ευρωβουλευτής πριν για την προηγούμενη αναφορά είπε τι θα κάνουμε και νομίζω αυτό θέλει και ο αναφέρον. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τη συμμόρφωση. Δεν μπορούμε να την επιτύχουμε 100% αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και το πρώτο βήμα είναι να ε, πιέσουμε την Ισπανία το ταχύτερο δυνατόν να υιοθετήσει αυτά τα προγράμματα διαχείρισης των λεκανών απορροής. Τα σχέδια τώρα είναι στο στάδιο των διαβουλεύσεων και θα συνεχίσουν μέχρι 27 Σεπτεμβρίου να είναι αντικείμενο διαβουλεύσεων. Η Ισπανία έδωσε κάποιες ενδείξεις ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα εγκρίνει όλα τα προγράμματα, αυτά τα σχέδια, θα δούμε, θα παρακολουθούμε, αλλά τώρα για να εγκριθούν τα μέτρα και να εφαρμόζονται αυτό θα γίνει. Θα αρχίσει η διαδικασία αξιολόγηση για να δούμε αν υπάρχει παραβίαση της οδηγίας ή όχι. Στην προηγούμενη αναφορά ακούσαμε διστάμενε απόψει από ανθρώπου που γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από μένα που είμαι νομικό, γιατί αυτό είναι τεχνικό θέμα και ίσω κάποιο ε, ειδικό στα τεχνικά, τεχνολογικά πρέπει να έρθει. Αλλά βλέπω διστάμενε απόψει. γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην μπούμε οριστικά αν υπάρχει παραβίαση της οδηγία ή όχι. Αν παραβιαστεί, ό,τι αφορά την εφαρμογή στο εθνικό επίπεδο. Ε, μπορεί να μην δόθηκε το σχέδιο μέχρι την τάδη ημερομηνία, θα πάει στην, ε, στο δικαστήριο και θα κρίνει. Αλλά όταν μιλάμε για οικολογικά θέματα, ροές, κίτες κλπ, εκεί είναι διαφορετικό. Πρέπει λοιπόν να δούμε πότε θα εγκριθούν και θα κοινοποιηθούν στην Κομισιόν. Είναι μακρά διαδικασία τα ε, σχέδια. Δεν θα μιλήσω με την, θα μιλήσω με με την Ισπανία τώρα Έχουμε ας πούμε με την ε, Ρουμανία διμερείς ε, συνομιλίες. Θα περάσουμε από αυτό το στάδιο και τότε ο αναφέρον, αν θέλει να επηρεάσει περισσότερο τη διαδικασία, μπορεί να υποβάλει σχόλια πάνω σε αυτά τα σχέδια και θα δούμε, θα τα συζητήσουμε, θα δούμε τι θα τα κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι θα την πάμε στα δικαστήρια την Ισπανία, αλλά μπορεί να πιέσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση μαζί με εσά για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όπως είπε σωστά και ο κύριος Ευρωβουλευτής, με βάση τους περιορισμούς από την νομοθεσία. Ελπίζω να απάντησα, ήμουν όσο σαφέστερος γινόταν σε αυτό το στάδιο. Anybody want to Άλλος, ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες. Ευχαριστώ. Θέλω να χαιρετήσω τους αναφέροντες που είναι συντοπίτες μου και θέλω να σας πω ότι από το 77 ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Σε αυτό το κουρμπέτι είμαι. 22 χρόνια βουλευτή στην επαρχία της Ciudad Real την οποία αφορά άμεσα το θέμα, όπως γνωρίζετε, και 14 χρόνια θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας χαιρετίζω λοιπόν, σας λέω ότι το πρόβλημά σας και η ανησυχία σας είναι αδιαφυσβήτητα κάτι που ε, συμμερίζεται σύσσωμος ο πληθυσμός της Καστήλης Λαμάντσα, τουλάχιστον στις επαρχίες της αυτόνομης αυτής κοινότητας, όπου ο ποταμός Τάχο ε, αποτελεί και τη σπονδυλική τους στήλη. Ε, είναι σαφές ότι σας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει το θέμα, το οποίο ε, προκάλεσε και μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Η πολιτική του νερού ε, παραμένει ανοιχτή, είναι ένας αγώνας που δίδεται κάθε μέρα. Θέλουμε αυτή η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή με το ίδιο πνεύμα υπό το οποίο διατηρήσαμε ανοιχτή την προηγούμενη αναφορά. Εγώ τρέφω ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς τα θέματα αυτά και πολύ συχνά υπάρχει σύγχυση για το ποιο είναι το καθήκον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποιο είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μόνη εξουσία που έχει η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να μελετήσει προσεκτικά τις καταγγελίες των πολιτών ή των συλλογικοτήτων των πολιτών για να διαπιστώσει εάν ε, εφαρμόζονται ή όχι οι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, οι ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις. Δεν μπορούμε ως Επιτροπή να επικρίνουμε ε, και να αποφανθούμε ε, περί μελλοντικών σχεδίων. Και πολύ συχνά οι πολίτες απογοητεύονται, γιατί νόμιζαν ότι θα έρθουν εδώ και ε, θα τους υποστηρίξουμε μέχρι τέλους. Αλλά είναι εκτός των καθηκόντων μας αυτό. Δεν μπορούμε να αποφαθούμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις προθέσεις και τη βούληση και τα σχέδια της εκάστοτε κυβέρνησης ή του οποιοδήποτε. Δεν μπορούμε ως Επιτροπή να σχολιάσουμε πολιτικές που θα εφαρμοστούν κάποια στιγμή στα κράτη-μέλη. Να κρίνουμε σχέδια και εφαρμογές που έχουν ήδη ξεκινήσει, που δρομολογούνται, που εφαρμόζονται και να πούμε κατά πόσο συνάδουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή όχι αυτές οι, αυτά τα καλέσματα, οι εκκλήσεις ε, για να εφιστήσουμε την προσοχή είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και να μην νομίζετε εσείς οι πολίτες ότι θα ανακαλύψουμε καταστάσεις που δεν έχουν ήδη καταγγελθεί, που δεν έχουν ήδη χαρακτηριστεί ή που δεν έχουν ήδη εκφραστεί. Είναι πράγματα που ήδη έχουμε κάνει. Και σε άλλες επιτροπές ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για παράδειγμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νομοθετική, νομοπαρασκευαστική ευθύνη, όχι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Αναφορών. Και εκεί είναι που διαμορφώνονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τις οποίες μιλούμε. Είναι οδηγίες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που πολύ συχνά εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και το Συμβούλιο ενδεχομένως καθιστούν εφικτή τη σύνταξη νομοθεσίας η οποία μας επιτρέπει να παρέμβουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις όταν διαπιστώνουμε τέτοιου είδους καταστάσεις και προβλήματα. Θέλω να εκφράσω την ελεγγύη μου, τη στήριξή μου ε, όλων μας. Είναι απόλυτα δικαιωμένη. Είναι θλιβερή η εικόνα που βλέπουμε στην οθόνη. Και οι εικόνες που δείξατε δεν είναι και οι πιο δραματικές. Υπάρχουν εικόνες πολύ πιο δραματικές. Ε, εμένα μου σηκώνονται τα μαλλιά όρθια κάθε φορά που το λέω, κάθε φορά που το ε, σκέφτομαι. παρακαλώ κυρία Πρόεδρε να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή να συνεχίσουμε να ανημερώνομαστε, να συνεχίσουμε να πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών οι οποίοι απευθύνονται σε εμάς και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί να μην υπερβάλλουμε για το πεδίο της αρμοδιότητας, της εξουσίας και της ικανότητάς μας. Ευχαριστώ ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή, όχι μόνο γιατί είναι σημαντική, αλλά γιατί είναι σημαντικό να γίνει η συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που να ξεπερνά αυτόν τον ποταμό. Πρέπει να κάνουμε μια τεράστια συζήτηση για τους υδάτινους πόρους. Δεν είναι τοπικό αυτό το θέμα, είναι παγκόσμιο, είναι συνολικό, είναι γενικό. Έχουμε πολιτική ευθύνη να μην το κλείσουμε και να μην... Ε, παραγνωρίσουμε την ε, συνολική διάσταση του προβλήματος των υδάτινων πόρων. Έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε σε φάση προσχεδίου αυτή τη στιγμή. Όμως συμφωνώ και με τον κύριο Μαρτίνεθ. Άλλο πράγμα η κινητοποίηση και άλλο η συμμετοχή σε μια διαδικασία. Έχει υπάρξει πολλή κινητοποίηση και θα υπάρξει και καλώς υπάρχει. Αλλά το ότι κινητοποιείται ο κόσμος δεν σημαίνει ότι συμμετέχει εξίσου μαζικά στην διαδικασία. Και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βούληση αυτή η κινητοποίηση να μετατραπεί σε συμμετοχή στη διαδικασία. Και ως Επιτροπή Αναφορών νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Η δουλειά μας είναι να τους προσφέρουμε αυτό το χώρο ώστε την κινητοποίηση να τη μεταφράσουν σε συμμετοχή στην διαδικασία. Δεν μιλούμε μόνο για ένα περιβαλλοντικό και οικολογικό πρόβλημα. Μιλούμε κατά κύριο λόγο ε, για οικονομικούς δεσμούς και ενδεχομένως διαπλοκές. Το οξύ πρόβλημα ε, που θα δημιουργηθεί εάν δεν δράσουμε πολιτικά εγκαίρως είναι το αναντίστρεπτο, ο αναντίστρεπτος χαρακτήρας. Εάν προκληθεί η βλάβη δεν υπάρχει σημείο επιστροφής. Είναι αδύνατο να επανέλθουμε στην, πρότερα, στην προτέρα κατάσταση και γι' αυτό πρέπει να δράσουμε εκ των προτέρων. Όχι μόνο ε, να μην ε, τεμπελιάσουμε αν θέλετε και να μην ε, επαναπαυθούμε αλλά να αντλήσουμε και τα διδάγματα του παρελθόντος. Ξέρουμε ορισμένες ε, ε πολιτικές ομιλίες, ορισμένοι πολιτικοί λόγοι, ευχολόγια και διακηρύξεις που μας έχουν οδηγήσει στο παρελθόν δεν πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα ε, μόνο από την πλευρά των τοπικών συμφερόντων ή ενδιαφερόντων, αν θέλετε, του τοπικού πληθυσμού. Είναι ένα θέμα με παγκόσμιες, με συνολικές προεκτάσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέγερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την πλατφόρμα υπεράσπισης του ποταμού Τάχου, αλλά και τον συντονιστή της Ενωμένης Πράγματι, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της οδηγίας, η μερική εφαρμογή της οδηγίας υποχρεώνει την ε, οργανωμένη κοινωνία των πολιτών να αντιδράσει, να αντιδράσει σωστά και εγκαίρως. Είναι, είναι καλό λοιπόν που γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα πριν υπάρξει οριστική έγκριση του σχεδίου. Ο ποταμός Τάχο και ο ποταμός Σεγούρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη λόγω της πολιτικής των φραγμάτων και εκτροπών. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις λεκάνες απορροής. Πράγματι η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. 15 κυβικά εκατοστά για τον Τάχο και 5 ε, κυβικά εκατοστά για το Αλμπέρτσε είναι ε, μια τεχνική προϋπόθεση για τη διατήρηση του οικολογικού ε, διάβλου και κήτης, αν θέλετε, των ποταμών. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ θα θέσω στους συντονιστές το εξής. Να, αν επισκεφθούμε το δέλτα του Εύρου, να επισκεφθούμε και το ποτάμι Τάχο. Ξέρω ότι έχουμε πολύ περίπλοκο χρονοδιάγραμμα. Αλλά νομίζω ότι είναι εφικτό ε, να καταφέρουμε να επισκεφθούμε και τα δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θέλουν να δευτερολογήσουν για ένα λεπτό οι, ε, ε, αναφέροντες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την Επιτροπή Αναφορών για την υποδοχή που μας επιφύλαξε, για το ότι μας άκουσε, για το ότι είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να εργάζεται πάνω στην εξέταση αυτής της αναφοράς για το ότι θέλει να τη διατηρήσει ανοιχτή την αναφορά αυτή. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ε, η κατάσταση του ποταμού ε, Τάχο είναι πραγματική. Βλέπετε τη φωτογραφία. Έτσι είναι η κατάσταση εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Μακάρι να μπορούσατε να πάτε στο Τολέδο και στην Ταλαβέδα Τε Λαρέινα και να δείτε πώς είναι τα χέλια π.χ. στο ποτάμι. Αν τον δείτε από κοντά θα εκπλαγείτε με την κατάσταση. Είναι ισπανικό ποτάμι, ανήκει σε όλους, αλλά πρώτα απ' όλα είναι ποτάμι και αυτή τη στιγμή δεν είναι. Πρέπει να το ανακτήσουμε και να το ξαναδημιουργήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που καταδείξατε τα σημαντικότατα αυτά ζητήματα. Παραμένει ανοιχτή η αναφορά γιατί πρέπει να δούμε ποιες είναι οι μελλοντικές εξελίξεις. Ελπίζουμε μέχρι τα τέλη του έτους να έχουμε θετικά νέα. Επομένως, διατηρούμε ανοιχτή την αναφορά και θα συνεχίσουμε την όλη εργασία της παρακολούθησης υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Μαδρίτη και για την έκθεση αυτή δίνω το λόγο στην κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχαμε στείλει στην Μαδρίτη μία αντιπροσωπεία 21-22 Μαρτίου να, στα πλαίσια του νομοθεσίας για τις ακτές. Η μερίσια διάταξη είναι γνωστή. Θέλω να πω ότι υπήρχε μεγάλη συμφωνία μεταξύ των μελών ότι ήταν καλή η συνεργασία μεταξύ των τακτικών μελών και των μελών εξοφίτσιο και με τη γραμματεία. Ε, τα μέλη εξοφίτσιο ήταν ε, πολύ καλά ενταγμένα στην ομάδα, το επιβεβαιώνει νομίζω και ο συνάδελφος Γιάρ. Το έγγραφο το έχουμε. Το Σεπτέμβριο θα έπρεπε να υποβληθούν οι τροπολογίες, πρέπει να υποβληθούν οι τροπολογίες και το έγγραφο αυτό θα είναι κομμάτι της ομάδας εργασίας στην ίδια την ομάδα εργασίας όμως θέλουμε μια συνάντηση ακόμα στις αρχές Σεπτεμβρίου για να αποφασίσουμε τα περαιτέρω της ομάδας αυτής και θα συζητήσουμε και την έκθεση και πάνω απ' όλα τις τροπολογίες. Νομίζω ότι η, η συνέχεια που δόθηκε στις αναφορές ε, εξηγούνται καλά στην έκθεση και οι ε, συνομιλίες με τους αναφέροντες και τους άλλους ε, ενδιαφερόμενους. Όλα ε, αντικατοπτρίζονται καλά. Καλά παρατηθένται συναντήσεις, συναντήσεις με τους αρμόδιους. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ, αυτά είχα να πω από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω πρέπει να λάβει το λόγο. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά στην έκθεση αυτή μετά την επίσκεψη και εμείς εκ του σύνεγγης παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, στο δικαιικό σύστημα της Ισπανίας. Είπαμε δεν υπάρχουν ε, ιδιαίτερες αρμοδιότητες για παρέμβαση με βάση το νοσιακό δίκαιο, αλλά επειδή είναι σημαντικό το θέμα και πολύ ενδιαφερόμενοι παρακολουθούμε από κοντά και θα συνεχίσουμε βέβαια να παρακολουθούμε την εξέλιξη του νομικού πλαισίου στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρίσο Μαρτέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι από περιβαλλοντική σκοπιά η κατάσταση είναι περίπλοκη. Πολλά είναι τα στοιχεία, οι πληροφορίες. Θα παρακολουθήσουμε στενά την αυστηρή εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θα κάνω μια πολιτική εκτίμηση, γιατί έχουμε διαφορετική άποψη σε σχέση με την Κομισιόν. Η διαρνητική επίστο... Ε, ναι, επίσκεψη μας απέδειξε ότι έπρεπε να δούμε στη Μαδρίτη και τους κυβερνητικούς εκπροσώπους και τους αναφέροντες, γιατί πρόκειται και για περιουσιακά δικαιώματα πέρα από το περιβάλλον, ε, θα πρέπει η ελευθερία της αγοράς να προστατεύεται και στο μέλλον. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό γιατί είναι δίκαιο στην Ευρώπη και είναι θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών. Γι' αυτό στην Επιτροπή Αναφορών ασχοληθήκαμε ε, αντίθετα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιβεβαιώθηκα στις αρχικές μου εκτιμήσεις. Δεν είμαι νομικός, μιλώ εδώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήθελα καταρχήν να μιλήσω θετικά και να επενέσω τη γραμματεία. Αυτή ήταν μια στενά οριοθετημένη και πολύ αποτελεσματική διερευνητική αποστολή που λειτουργήσε εξαιρετικά γιατί πάντοτε είναι επικίνδυνο, υπάρχει ο κίνδυνος να νιώσει κανείς ανία, πράγμα που δεν συνέβη καθόλου ε, στην αποστολή μας αυτή. Επίσης θέλω να επενέσω και την επικεφαλής της αντιπροσωπείας, γιατί εδώ ε, βρήκα μια συμβαστική λύση σε σχέση με το ταξίδι και ομόφωνα συμφωνήσαμε σχετικά με αυτά που είδαμε. Ε, είναι σημαντικό να υπάρχει συνένεση. Η κυρία Βέρτμαν ε, έλαβε υπόψη της και τα ε, εξοφίτσιο μέλη τους Ισπανούς συναδέλφους και ήθελε να τους εντάξει στην αποστολή για να συμβάλλουν και εκείνοι σε μια λειτουργική συμβιβαστική λύση. Νομίζω ότι μπορούμε να ε, παρουσιάσουμε και κάποια αποτελέσματα. Α, και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι πρέπει να επενεθούν. Γιατί όταν μιλήσαμε για την Κοπενχάγη θα δούμε ότι δεν είναι αυτονόητα όλα αυτά. Στην Ισπανία, τη Μαδρίτη, είχαμε ανοίχ τη ατμόσφαιρα επικοδομητικού διαλόγου και υπήρξαν και βελτιώσεις. Υπήρξε τώρα νέος νόμος για την προστασία των ακτών στην Ισπανία και νομίζω ε, ότι και αυτά πρέπει να τα πούμε εκτός από τις κριτικές παρατηρήσεις που έχουμε. Βέβαια δεν πρόκειται μόνο για προστασία του περιβάλλοντος εδώ, αλλά πρόκειται και για το δικαίωμα απόκτησης περιουσίας και τα περιουσιακά δικαιώματα. Τώρα, όταν δούμε τα έγγραφα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο νόμος για την προστασία των ακτών στην Ισπανία αναθεωρήθηκε, τροποποιήθηκε και θα πρέπει να δούμε το περιεχόμενο του νέου νόμου για την προστασία των ακτών και να το συμπεριλάβουμε στην εκθεσή μας, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε σε ποιο σημείο του εγγράφου μας θα το εντάξουμε και αυτό. Για μένα το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να δούμε το πρόβλημα των δικαιωμάτων ε, της ιδιοκτησίας. Πρέπει να παρακαλέσω με τις ισπανικές αρχές να φροντίσουν να βρεθεί ένας, ε, μια νομική οδός αποτελεσματική σχετικά με το πού θα ε, ε γύρει τις αξιώσεις του ένας πολίτης. Ε, είδαμε δύο ακραίες καταστάσεις, ένας ε, αγρότης είχε από την εποχή του Κολόμβου ένα αγρόκτημα και θα έπρεπε να ε, φύγει από εκεί για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Ε, μετά έχουμε και κτίρια γραφείων τα οποία κατασκευάστηκαν στην ακτή και προστατεύονται τώρα. Ε, πάντως, ναι, γι' αυτό λέω ότι ήταν μια πολύ κατατοπιστική διερευνητική αποστολή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικά αυτά που είδαμε. Η κυρία Άουκεν. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Γραμματεία, την Αγγέλικα επίσης, η οποία μέχρι στιγμής κινήθηκε τουλάχιστον πολύ ομαλά στη συνεργασία που είχαμε και είχαν γίνει βέβαια κάποιες απόπειρε στην αρχή η Επιτροπή μας αυτή να μην έχει αρκετά μεγάλη πυγμή και να μην προσβάλλουμε καμία αρχή, ιδίως να αυτή προέρχεται από ένα από τα μεγάλα κόμματα. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό καθιστά τα πράγματα πολύ δύσκολα. Γιατί όταν ταξιδεύουμε και προσπαθούμε ουσιαστικά να εκπροσωπήσουμε τους αναφέροντες, των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται, Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε, τι λέμε και τι βλέπουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η μάχη αυτή την οποία δίνουμε είναι μία μάχη που δίνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν εγκρίθηκε η έκθεση μου το 2009 από την Ολομέλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει τότε ότι θα ασχολείται με τα ζητήματα αυτά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε είχε πει ότι εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε πραγματικά να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό και ότι αποτελεί και αυτό δική μα αρμοδιότητα. Βέβαια, τα πράγματα είναι κάπω πιο δύσκολα και διαφορετικά όσον αφορά το δίκαιο για τι παράκτη περιοχέ τη Ισπανία, γιατί ουσιαστικά καλύπτει πολλέ διαφορετικέ οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση την έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου μα λέει ότι δεν είναι αρμοδιότητά του. Τουλάχιστον πέντε οδηγίε εμπίπτουν σε αυτό το εθνικό δίκαιο για τις παράκτης περιοχές Ισπανίας. Και βέβαια παράλληλα υπάρχει και τώρα το ζήτημα του διοκτησιακού καθεστώτος. Όσον αφορά κάποια συμπεράσματα και κάποιες συστάσεις, αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν βελτιώθηκε η νομοθεσία με τον νέο αυτό νόμο. Έχουμε ουσιαστικά ένα νέο νόμο, ο οποίος ε, σε σχέση με το παλιό δεν εφαρμόζεται. Ο παλιό νόμο τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ καλό για το περιβάλλον, αλλά τουλάχιστον εφαρμοζόταν. Ο νέο νόμο τη Ισπανία δεν είναι θετικό για το περιβάλλον, δεν είναι φιλικό προ το περιβάλλον και δημιουργεί πάρα πολλέ ε, συγχύσει και αμφιβολίε όσον αφορά το ειδικτωσιακό καθεστώ, όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησία των πολιτών. Θεωρώ ότι λειτουργεί με τρόπο ιδιαίτερα αυθαίρετο και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι προστατεύονται τελικά μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις ξία. Βλέπουμε ότι έχει έρθει αυτή η νέα ισπανική νομοθεσία, η οποία ουσιαστικά υποφελεί περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα που είχαμε με την παλαιότερη νομοθεσία ήταν ότι δεν εφαρμοζόταν βέβαια. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα κινηθούν θετικά και ότι μετά την επίσκεψη αυτή και μετά από τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει, τα πράγματα θα κινηθούν καλύτερα για το ζήτημα του δικαίου για τις παράκτη περιοχές. Ο κύριος Βίλαντ. Μάλλον ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο νόμος για τις παράκτιες περιοχές ήταν ένας νόμος τον οποίο πρότεινε και ενέκρινε ε, το Ισπανικό Κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας κυβέρνησης του δικού μου κόμματος. Ήταν, είχε καλές προθέσεις ο νόμος αυτός και προφανώς δημιούργησε πολλά προβλήματα. Δεν το αφιζητώ αυτό. Διότι απόδειξη αυτού είναι ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός των αναφορών που μας υποβλήθηκαν και που σχετίζονται με την εφαρμογή δεν συμφωνώ με την κυρία Άουκεν, η οποία δεν με ακούει και συνηθίζει να μην με ακούει. Εφαρμόστηκε, κυρία Άουκεν, ο νόμος τόσο πολύ που υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές λόγω της εφαρμογής του νόμου αυτού. Ήταν καλός αυτός ο νόμος κατά τη γνώμη μου, ωστόσο αυτό που ε, κατέδειξε είναι ότι είναι εφιαλτικά περίπλοκο το θέμα αυτό και συμφωνώ με την κυρία Άουκεν στο ότι δεν εφαρμόστηκε πάντοτε με τον πιο έξυπνο τρόπο ο νόμος αυτός και δεν εφαρμόστηκε λαμβάνοντας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συμφέροντα που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Ενεκρίθη με ενθουσιασμό από τις οικολογικές οργανώσεις που είχαν συμμετάσχει στην Παρασκευή αυτού του νόμου και η κυβέρνησή μας τον ψήφισε μεριμνώντας ιδιαίτερος για, τον περιβάλλον, για το περιβάλλον, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι αυτός ο νόμος θα έπλητε άλλα συμφέροντα. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που δημιούργησε ο νόμος και τις παζοκεφαλιές που ε, δημιούργησε τελικά για ορισμένους από εμάς. Είναι λογικό αυτό που είπατε, είναι λογικό και η παρουσίαση της συναδέλφου. Λυπούμε που δεν υπάρχει κανείς συμπατριώτης μου αυτή τη στιγμή από το Λαϊκό Κόμμα εδώ για να σχολιάσει, να πει την άποψή του, να ε, παρεύει με τρόπο που δεν μπορώ να ε, παρεύω εγώ. Το μόνο που θέλω να πω στην κυρία Άουκεν είναι το εξής. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στον νόμο έγιναν μόνο και μόνο επειδή οι οικολογικές οργανώσεις ήταν εναντίον της μεταρρύθμισης. Η κυρία Άουκεν έχει θέμα με την ιδιοκτησία. Εγώ δεν είμαι παδός του Σιλίπ Χουντόμ που έλεγε ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή. Πιστεύουμε όμως ότι υπερισχύει η υπεράσπιση της φύσης του περιβάλλοντος, του κόσμου. Για άλλους ε, το πρωταρχικό είναι η ιδιοκτησία και ότι αυτό είναι ε, μια ιερή αγελάδα ε, που πρέπει οπωσδήποτε να σεβαστούμε. Το σημείο ισορροπίας είναι το θέμα μεταξύ των δύο. Αναρωτιέμαι, μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία σε τέτοια θέματα. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο, που ασχολούνται με το θέμα αυτό όχι μόνο γιατί ε, ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά γιατί ενδιαφέρονται και για ένα πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή πώς θα φτάσουμε σε σημείο, σε ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του γενικού συμφέροντος, που είναι δηλαδή η προστασία των παράκτιων περιοχών και της προστασίας της ιδιοκτησίας και των ιδιωτικών συμφερόντων. 72 εκατομμύρια τουρίστες θα έχουμε του χρόνου, για παράδειγμα, κυρία Πρόεδρε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σειραίουν στις ισπανικές ακτές, οι οποίες έχουν υποφέρει πάρα πολύ. Βεβαίως έχουν αναπτυχθεί άνευ προηγουμένου, αλλά έχουμε τεράστιες ανισορροπίες, τεράστιε διαφορές είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται, πρέπει να εφαρμόζονται και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για να συγκεραστούν όλα τα συμφέροντα. Εμείς επανειλημμένως έχουμε συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σήμερα από ό,τι υπήρχε εδώ και 40 χρόνια για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Και προς το συμφέρον του τουρισμού είναι αυτό. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος βοηθάει στον τουρισμό. Όταν καταστρέφεται το περιβάλλον είναι σαν να σκοτώνουμε ακριβώς αυτή την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη στήριξή τους, για για την βοήθειά τους κάθε φορά που υπήρξε καταγγελία, κάθε φορά που υπήρξε αίτημα για βελτιώσεις. Πάντοτε με σεβασμό, χωρίς εχθρικότητα, χωρίς εχθρικό πνεύμα ούτε εναντίον της Ισπανίας ούτε εναντίον της Επιτροπής. Το μόνο που θέλουμε όλοι είναι το καλύτερο δυνατό για όλους. Ευχαριστώ κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι όλους και τα τακτικά και τα εξοφίτσιο μέλη και θέλω να αναφέρω πολύ θετικά την καλή συνεργασία που είχαμε στην Ισπανία με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης γιατί συμφωνώ με τον Πέτερ μάθαμε στην επίσκεψη ότι και από, τη, από άλλες επισκέψεις ότι αυτά δεν είναι δεδομένα πάντοτε. Οπότε τα σημειώνω πολύ θετικά. Πρέπει επίσης να διαβεβαιώσω όλους τους Ισπανούς συναδέλφους ότι γνωρίζομαι πολύ καλά πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα. Ε, δύσκολα, ε, πολλές φορές τα καταλαβαίνουμε, καμιά φορά και όταν μιλούσαμε με τους αναφέροντες και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ε, ε, είχαμε κάποιες δυσκολίες κατανόησης, το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και με τον απαιτή σεβασμό προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε. Κάνουμε μεγάλες και σκληρές προσπάθειες. Γι' αυτό, ε, όπως ο Πέτερ, ε, καταλήξαμε σε συνένεση ο Πέτερ προτείνει να αναφερθούμε και στον νέο νόμο. Ε, δεν θα το αποφασίσω βέβαια αυτό εγώ, αν θα το συμπεριλάβουμε στην έκθεση ή όχι. Πρέπει να συζητήσουν τα τακτικά μέλη για το θέμα ή να το θέσουμε στην ομάδα εργασίας στην συνάντηση του Σεπτεμβρίου και να το συζητήσουμε εκεί, γιατί είναι αυτό ένα σχόλιο, είναι ένα θέμα που πρέπει και αυτό να συνεξεταστεί. Από την πλευρά μου ελπίζω ότι θα μάθουμε γρήγορα μέχρι πότε θα μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες στις συστάσεις ώστε να συμπεριληφθούν και να συμμετέχουν στη διαδικασία όλα τα μέλη της Επιτροπής και τέλος άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Όλους σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε την έκθεση τον Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ, είμαι πολύ ικανοποιημένη που μπορούμε να καταγράψουμε αυτή τη συνένεση. Ευχαριστώ όλους. Προχωρούμε τώρα. Στην επόμενη έκθεση από την διερευνητική επίσκεψη στη Δανία και δίνω το λόγο πάλι στην κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας που στις 20 και 21 Ιουνίου μας, πήγε στην, μας έφερε στην Κοπενχάγη. Ο Πέτερ Γιάρ και ο Κάλατι Κουργκάης ήταν το δεύτερο και το τρίτο μέλος μας. Εμείς πήγαμε εκεί σχετικά με τις αναφορές του Φεβρουαρίου που, αναφο... αφορούσαν δικαιώματα παιδιών, διακρίσεις σε βάρος των γονέων και διακρίσεις σε βάρος των μητέρων στη Δανία. Μετά από τις συζητήσεις του Φεβρουαρίου λοιπόν, πολλές ακόμη αναφορές παρελήφθησαν από την Επιτροπή. Τώρα αξιολογούνται. Νομίζω ότι πρέπει να παρουσιάσουμε κάποια σχόλια από την εμπειρία μας στην Δανία. Ζητήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δυστυχώς και οι δύο υπουργοί μας εγνώρισαν ότι δεν μπορούσαν να μας συναντήσουν, παραθέτω, διότι, ε, διότι είχα, ήταν στις θερινές διακοπές. Τέλος του παραθέματος. Ε, οι υπουργοί αρνήθηκαν μία συνάντηση επίσημη ε, με μία επιτροπή που έχει λόγο στα θέματα αυτά μέσα στο Κοινοβούλιο. Πρώτη φορά μου συνέβη κάτι τέτοιο. Και βεβαίως ε, ανησυχώ πάρα πολύ. Προσωπικά συμπεραίνω από την απόρριψη αυτή μια συνάντησης με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε επίσημη αντιπροσωπεία είναι ότι αυτό η απόρριψη δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα πολιτικό και όντως το πρόβλημα είναι σοβαρότερο από ό,τι μπορούμε να κρίνουμε αυτή τη στιγμή και θα το εξηγήσω και αργότερα αυτό. Ε, μαθα επίσης ότι ο Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων δυστυχώς κοινοποίησε στη Δανία ότι, στην κοινή γνώμη ότι εμείς δεν θέλαμε να ε, τον δούμε και να δούμε εκπροσώπους του και δεν θέλαμε να συζητήσουμε λεπτομέρειες. Η υπουργό είναι η γυναίκα. Και είπε ότι θέλαμε εμείς να συζητήσουμε πολύ λεπτομερή θέματα. Εμείς και οι τρεις είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και για λεπτομέρειες και κάναμε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα τα ίδια. Δυστυχώς οι εκπρόσωποι με τους οποίους μπορέσαμε να μιλήσουμε, είτε ήταν η Υπουργό ε, Κοινωνικών Υποθέσεων ή Υπουργό Δικαιοσύνη, κάποιοι από το γραφείο των Υπουργών δεν ήταν προετοιμασμένοι και καμιά φορά αρνήθηκαν να μας απαντήσουν και αυτό μας έκανε να συμπεράνουμε δυστυχώς ότι έπρεπε να γυρίσουμε στις Βρυξέλλες με πολύ περισσότερες ερωτήσεις από ότι όταν ξεκινήσαμε. Επίσης ο τρίτος ε, αξιωματούχος, τρίτος στη τάξη ήταν ο επικεφαλής της Δανική Αστυνομίας. Δυστυχώς και αυτός ε, έστειλε μέλη από το γραφείο του, δεν ξέρω ε, πώς, ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί, κάποιοι συνεργάτες, κάποιοι ειδικοί ήρθαν, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν. Δεν ήταν έτοιμοι να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι όλους πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα και τι συνέπειες έχει και τι πρέπει να πούμε. Το βράδυ της Πέμπτης είδαμε τους αναφέροντες και ανθρώπους που ήδη είχαν υποβάλει μια αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών, τη δική μας εδώ στο Κοινοβούλιο και συναντήσαμε επίσης και άλλους ανθρώπους που, στην ίδια συνάντηση που επρόκειτο να υποβάλουν αναφορά. Ήταν πάνω από 35-40 άνθρωποι παρόντες, μητέρες, πατέρες, εκπρόσωποι ε, των ανησυχούντων γονέων. Η συνάντηση διήρκεσε για περισσότερες από τέσσερις ώρες χωρίς διακοπή. Πρωτοφανές, κανείς από τους τρεις μας, συμπεριλαμβανώντας και τον κύριο Χέσεν από τη Γραμματεία, δεν ε, έφυγαν, διότι αυτές οι ιστορίες συνάδελφοι ήταν πολύ συγκινητικές πράγματι. Μάθαμε για σωματική βία ε, από γονείς σε παιδιά και σεξουαλική βία σε βάρος πολύ μικρών παιδιών. Αυτά τα παιδιά κάποιες φορές ερωτήθηκαν από το σχολείο ή τον νηπιαγωγείο και τα, μέσα ε, ανάκρισης των παιδιών τα αποτελέσματα από τις ανακρίσεις παρουσιάστηκαν στους ε, ενόχους γονείς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το παιδί. Πρέπει να, το παιδί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Φανταστείτε πώς νιώθει το παιδί ότι εμπιστεύεται σε κάποιον ε, ε, εμπιστεύεται κάποιον και του λέει τι συνέβη και μετά όλα αυτά τα ακούει ο πατέρας, αυτό είναι κατανοητό γιατί πρέπει να ερωτηθούν και οι γονείς, ο πατέρας, Και βέβαια μετά είπαν ότι όλα είναι εντάξει, το παιδί μου λέει ψέματα, είπαν οι γονείς. Αυτό το παιδί θα αναγκαστεί τότε να ξαναγυρίσει σε αυτόν τον πατέρα που ε, ασκηβία σε βάρος του. Και αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα μόνο στη Δανία. Αυτό είναι πρόβλημα σε οικογένειες άλλες ή οικογένειες τρίτων χωρών από την Αμερική ή την Ασία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας, πρέπει να μας εμπιστεύονται και γι' αυτό πρέπει εμείς να τους πάρουμε πολύ σοβαρά. Το επόμενο πρωινό συναντήσαμε τον συνήγορο του πολίτη. Δύο-τρία λεπτά δώστε μου ακόμα κυρία Πρόεδρε. Ο Κάρλος θα μπορούσε ίσως να συνοψίσει πολύ καλύτερα από μένα τη συνάντηση αυτή και τον ευχαριστώ για την παρουσία του εκεί και για ό,τι προσέφερε. Ε, ήταν σε μια είναι σε μια αντιπροσωπεία στο εξωτερικό δεν μπορούσε να είναι ο ίδιος. Οι τρεις μας πάντως, για να μην μακρηγορώ, ε, καταλήξαμε σε μια συνένεση αμέσως, συνένεση όπως αρέσει να λέει ο Πίτερ. Αποφασίσαμε να δουλέψουμε γρήγορα, χάρη, χάρη και στη συνεργασία με τον David Love και, την, και τον George Χέισεν από τη Γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας και όλη την υποστήριξη που μας δώσατε σε αυτό το σημαντικό θέμα. Εγώ προσωπικά έμαθα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε πολύ σοβαρά τα προβλήματα των παιδιών και εν προκειμένου πρέπει να πω ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Δανία. Αφορά γονείς και παιδιά που ζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συμπληρώσω μερικά σε αυτά που είπε η κυρία Βέρτμαν. Η μερίσια διάταξη ήταν καλή, προετοιμασμένη από τη γραμματεία. Η... Το ταξίδι είχε ιδιαιτερότητες. Το ένα είναι ότι είδαμε αρχές που θεωρούσαν ότι έχουν την καλύτερη νομοθεσία του κόσμου και ότι δεν χρειάζονται τροποποιήσεις και αλλαγές. Το κλίμα ήταν μια φιλική συγκατάβαση ε, φιλική ήταν αλλά δεν ε, άλλαζαν γνώμη ούτε κατά κεραία. Ε, εμείς είδαμε γενικά την κατάσταση, δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει μελήματα των πολιτών και θα πρέπει βέβαια να εξετάσουμε και συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλιώς δεν γίνεται. Ε, έμοιαζε λίγο, έτσι για να το πω, αστεϊζόμενο σε ένα ταξίδι ε, στη Μόσχα επί ψυχροπολεμικού κλίματος, όπου έλεγε μην ανακατεύεστε σε ξένες υποθέσεις εσωτερικές, να μην ανακατευόμαστε, δηλαδή ήταν ένα μήνυμα. Βέβαια η Δανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να ασχοληθούν με κάποια θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ε, κάτι μοναδικό που με στενοχώρησε. Κανείς από το Δανέζικο Κοινοβούλιο δεν βρήκε το χρόνο να έρθει να μας συναντήσει και να μας συνοδεύσει. γιατί θα μπορούσαν να έρθουν και να μας εξηγήσουν και κάποια πράγματα και επανέρχομαι στις διαβουλεύσεις ε, με τον ε, συνήγορο του πολίτη. Καλό ε, θα ήταν να έχουμε και άλλες παρόμοιες συναντήσεις γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε σχέση με τις διακρίσεις που δεν μας παρουσιάστηκαν. Μια άλλη ιδιαιτερότητα ήταν οι μακρές διαβουλεύσεις με τους αναφέροντες, είπε και η κυρία, το είπε και η κυρία Βέρτμαν και ε, δεν θέλαμε να διακόψουμε ούτε να φύγουμε γιατί ήταν τραγικά αυτά που ακούσαμε. Από τη, από τη δική μας την πλευρά ε, πρέπει να πω ότι είδαμε ότι εδώ υπάρχουν εγκληματικές δραστηριότητες ε, και το να μην αντιδράσουμε θα ήταν σαν να γινόμαστε συνεργοί. Ε, αυτά τα θέματα ε, θα έπρεπε να παραπεμφθούν στην εισαγγελία στη Δανία η οποία θα έπρεπε να παρακληθεί να ασχοληθεί δελεχέστερα με αυτά τα θέματα γιατί δεν πρόκειται εδώ για θέματα πολιτικά ούτε θέματα που αφορούν την ιδιοκτησία αλλά είναι θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν. Συγγνώμη, δεν ε, μπορούσα να συμμετέχω, αλλά πήγαινα στο νοσοκομείο τότε. Πρέπει να κάνω μια επέμβαση, επομένως δεν μπορούσα να έρθω. Προφανώς θα έπρεπε να είμαι εκεί, θα ήθελα να είμαι μαζί σας. Δύο πράγματα μόνο θα πω. Πρώτον, βλέπετε ότι η Επιτροπή μας παραμένει άγνωστη στη Δανία. Θα μου πείτε, δεν σας νοιάζει καθόλου γιατί δεν αφορά τη δική σας τη χώρα αλλά αυτό είναι το ζήτημα το οποίο εγώ αντιμετωπίζω συνεχώς στη Δανία. Ακόμα και στις εβδομαδιαίες επαφές που έχω στην χώρα μου, τους ανθρώπους εκεί, πρέπει κάθε φορά να αναφέρομαι και να εξηγώ στην Επιτροπή Αναφορών διεξοδικά, προσπαθώντας να εξηγήσω στους ανθρώπους τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή μας. Δεύτερον, κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το μάθατε, η Δανία μετά την, με το κοινοτικό δίκαιο για τα διαζύγια, η, έχει ένα opt-out για το δίκαιο αυτό η Δανία και προσπάθησε μάλιστα να πετύχει μία συμφωνία η οποία ουσιαστικά δεν έγινε δεκτή. Επομένως, πρέπει να σας πω ότι δεν υφίσταται λοιπόν πλέον το δίκαιο αυτό. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε την ομολογία του δικαστηρίου σε μια χώρα, την ομολογία του δικαστηρίου σε μια άλλη χώρα και δεν υπάρχει καμία μέση οδός, καμία δυνατότητα να συνδυαστούν αυτές τι ομολογίες. Αυτό εμείς προσπαθήσαμε να θίξουμε και λυπάμαι που πραγματικά δεν σας το εξήγησαν αυτό οι δανέζικέ αρχές ότι δεν υφίσταται το κοινοτικό αυτοδίκαιο και ότι έπειτα εφαρμόζεται η κοινοτική νομολογία ακριβώς επειδή η Δανία έχει ζητήσει ένα opt-out για το ζήτημα αυτό. Και να σας πω κάτι ακόμα. Λυπάμαι πραγματικά που δεν ήρθατε σε επαφή με εκπροσώπους της κυβέρνησης. Ένας εκπρόσωπος από την Υπουργείο Εξωτερικών ήρθε σε επαφή μαζί μου και ήταν ιδιαίτερα διαλλακτικός. Και η όλη οδηγία που δόθηκε από την Υπουργείο Εξωτερικών ήταν πραγματικά να δείξουν μια θετική στάση. Θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι ε, η 21η Ιουνίου στη Δανία, εσύ καταλαβαίνεις, αν φτάσετε το βράδυ της 21ης Ιουνίου, όπου ε, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εγκαταλείπουν την εργασία τους, ξαστικά πάνε να γιορτάσουν ακριβώς επειδή γιορτάζουν το θερινό ηλιοστάσιο και πίνουνε, όχι στη Σουηδία το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι η χρονική στιγμή της επίσκεψης δεν ήταν καλή. Πραγματικά λυπάμαι που δεν έρθες σε επαφή με Λυπάμαι που έγινε και όλη αυτή η σύγχυση όσον αφορά το προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα. Σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι είναι σφάλμα βέβαια της δικής μας επιτροπής. Απλώς ήθελα να τα πω όλα αυτά γιατί άκουσα μια πολύ επικριτική στάση από διάφορους συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε κυρία Όκεν. Είναι η πρώτη μόνο ανταλλαγή απόψεων που έχουμε για την έκθεση αυτή. Θα έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεση στην επόμενη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Γνωμοδότηση του κυρίου Τσίτσεστερ. Έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτη λοιπόν ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες στην γνωμοδότησή μου. Γνωμοδότηση την οποία εμείς συντάσσουμε για την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, η οποία είναι η καθήλυνα αρμόδια για το ζήτημα αυτό, τον καθορισμό των ενδρών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα τη διπλή έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είχα το χρόνο να διαβάσω και να αναλύσω με κάθε λεπτομέρεια όλες τις 164 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση μεγάλος αυτός αριθμός τροπολογιών και όλος περιέργως περίπου ένα 85% τροπολογιών αυτών προέρχονται από Γάλλους συντάκτες. Για ποιο λόγο άραγε. Προσβλέπω πάντως σε περαιτέρω ανάλυση των τροπολογιών αυτών με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να καταφέρω και εγώ με κάθε λεπτομέρεια να απαντήσω σε αυτές τις τροπολογίες. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία προκύπτουν από τις τροπολογίες. Ορισμένες τροπολογίες προσπαθούν πραγματικά να ταχθούν κατά της νομικής βάσης της αναφοράς ή του όλου του ζητήματος. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ προς αυτό είναι ότι έχουν δοθεί ήδη κάποιες απαντήσεις στις καταγγελίες αυτές, αλλά ακόμα και για αυτούς που δεν αρέσκονται στο να συζητούν το ζήτημα αυτό ή που δεν θέλουν να τίθεται καν το ζήτημα αυτό, πρέπει να σας πω ότι ακόμα και αν θα αυτή το ζήτημα αυτό δεν θα τους ωφελήσει γιατί το ζήτημα σίγουρα θα ανακύψει πάλι στο μέλλον και θα πρέπει να έχουμε κατά νου και μια σειρά ψηφοφοριών στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες ε, καταδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλά μέλη του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην τωρινή θητεία αλλά και σε πρότερες θητείες, οι οποίες σαφώς έχουν ταχθεί με απόλυτη σαφήνεια για το ζήτημα του Στρασβούργου και των δύο εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στα όσα λέγονται από νομικής πλευράς. Θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό για τους νομικούς αλλά και για μένα και φαντάζομαι θα καταφέρω να βελτιώσω και τα γαλλικά μου από όλη αυτή την προσπάθεια. Ένα-δύο σημεία τώρα έχουν προκύψει. Πρώτον, μου λένε ότι ενδεχομένω να έχει γίνει κάποιο σφάλμα όταν προτείνεται ότι η έδρα του Στρασβούργου επελέγει για λόγους συμφιλίωσης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας για ιστορικούς λόγους. Νομίζω ότι είναι λογική η πρόταση αυτή, αλλά μου υπόθηκε ότι ο αρχικός λόγος που συνεδρίασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ήταν μόνο και μόνο επειδή το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε μία αίθουσα εκεί όπου θα μπορούσε να συνεδριάσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και ότι ε, τελικά ήταν ε, το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης και η έδρα του στο Στρασβούργο αποτέλεσε τελικά το σύμβολο συμφιλίωσης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Και είχε επελεγεί για το Συμβούλιο της Ευρώπης συγκεκριμένα να τοποθετηθεί, να οικοδομηθεί κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Πρέπει να σας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνεδριάσει άλλωστε και στο Λουξεμβούργο, τουλάχιστον αυτό το έκανε πολύ συχνά στο παρελθόν. Και βέβαια συνεδριάζει, όπως το ξέρετε, και στις Βρυξέλλες, όταν βέβαια δεν πέφτει το ταβάνι. Βέβαια ξέρετε ότι τα γεγονότα αυτά της πτώσης της οροφής ε, δεν περιορίζεται μόνο στις Βρυξέλλες. Ανάλογα γεγονό είχαμε δει πρόσφατα και στο Στρασβούργο. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια αποκλειστικότητα προς αυτό ανάμεσα στις δύο έδρες. Ένα άλλο σημείο το οποίο τίθεται και το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς ως σημείο νομικής υφής είναι η παρούσα κατάσταση όπου ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει 12 φορές στο Στρασβούργο και ότι αυτό αποτελεί τμήμα των συνθήκων. Αυτό αληθεύει. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τους Γάλλους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ε, καταφέρει να εξασφαλίσουν τις συνεδράσεις αυτές κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για την έδρα του Κοινοβουλίου ούτε σημαίνει ότι εμεί που πρέπει σε τακτική βάση να ταξιδεύουμε προ το Στρασβούργο δεν μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μα. Αρκεί βέβαια να μην υπάρχουν απεργίε ή να μην υπάρχουν προβλήματα στη μετακίνησή μα αυτή. Μπορούμε λοιπόν εμεί ελεύθερα και έχουμε κάθε δικαίωμα να εκφραζόμαστε για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στη μετακίνηση αυτή. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει εμεί να σιωπήσουμε μόνο και μόνο επειδή οι συνθήκε μιλάνε για την έδρα αυτή και κατοχυρώνεται στη συνθήκη η έδρα του Στρασβούργου. Επίση, αλλαγέ θα μπορούσαν να γίνουν και στη συνθήκη. Βέβαια, στα πλαίσια τη ε, τελευταία συνθήκη, και ξέρετε ότι υπάρχουν πολλέ συνθήκε στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρξαν και πάρα πολλέ αλλαγέ συνθήκε, μένω είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οι συνθήκε και προβλέπεται ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προτείνει πλέον μία αλλαγή για τη συνθήκη. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να παρεμποδιστεί, παρεμποδιστεί με συγχωρείτε, η δυνατότητα αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα άλλο ζήτημα ίσονο σημασία που μου έχουν θίξει κάποιοι συνάδελφοι από το Συμβούλιο της Ευρώπης μου έχουν πει ότι η ίδια η πόλη του Στρασβούργου δεν μπορεί να φιλοξενήσει τόσους πολλούς εργαζόμενους κάθε φορά που συνεδριάζουν παράλληλα Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι αυτό συμβαίνει μερικές φορές, δύο-τρεις φορές το χρόνο, όταν συμπίπτουν οι δύο συνελεύσεις και στην περίπτωση αυτή πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολλοί που σειραίουμε στο Στρασβούργο και δεν καταφέρνουμε να βρούμε δωμάτια στα ξενοδοχεία και το καθεξής. Και όταν λέω όλοι εμείς, αναφέρομαι βέβαια στο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο βέβαια υπερέχει των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα λοιπόν αυτά πιστεύω ότι καταδεικνύουν ότι το επιχείρημα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό από οικονομική πλευρά για το Στρασβούργο, ενδεχομένως να είναι κάπως υπερβολικό. Καταλαβαίνω βέβαια ότι υπάρχουν κάποια αριθμητικά δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν την θετική οικονομική επίπτωση που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, αλλά αντίστοιχα δεδομένα υπάρχουν και για το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητηθούν, όλε οι πτυχέ του ζητήματο πρέπει να αναλυθούν. Και α μην ξεχνάμε ότι μία αναφορά κατατέθηκε το 2006, η οποία φέρει πολλέ υπογραφέ και η οποία έγινε αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρήθηκε παραδεκτή και είναι ακόμα ανοιχτή η κυρία Μάλμστρομ μάλιστα είχε υποβάλει την αναφορά αυτή, ιδιαίτερα γνωστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμεί εδώ πέρα πρέπει να αναλύουμε και να εξετάζουμε τις αναφορές και δεν θα πρέπει βέβαια να παραβλέψουμε και αυτή την αναφορά. Αυτά είχα να σας πω. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσίτσεστερ. Το λόγο για ένα λεπτό έχει η κυρία Τίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Τσίτσεστερ. Χαίρομαι που είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω το 1,3 εκατομμύρια πρόσωπα που υπέγραψαν στην αναφορά της Ήλια Μάλμστρομ και συμμετείχαν στην εκστρατεία για τη μία έδρα αυτούς εκπρόσωπο είναι πολύ σημαντικό να με αλλαγή του άρθρου 48, με βάση το άρθρο 48 αλλαγή στη συνθήκη. Είναι πονίδιστο ότι είμαστε το μόνο κοινοβούλιο που έχει περισσότερες έδρες, τρεις, και νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πολλά έχουμε πει για δαπάνες όλα αυτά τα χρόνια. 169 με 240 εκατομμύρια στοιχίζει αυτή η υπόθεση και δεν είναι οι τιμές ε, οι τρέχουσες του 2013. Τελειώνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και δεν μπορούμε να το αμελήσουμε. Ε, έχει περάσει και η ώρα. Είμαι η μόνη που ήμουν από τις αρχικές ε, υπογραφές, είχα βάλει αρχικά την υπογραφή μου στην αναφορά αυτή. Κύριος Μπουλάν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τώρα την γαλλική πλευρά στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τσίτσεστερ. Τον ευχαριστώ για την γνωμοδότησή του. Ωστόσο πιστεύω ότι βλέπει ότι εμεί παίξαμε το παιχνίδι. Αρχικά δεν θέλαμε μια έκθεση για αυτό το ζήτημα γιατί η έκθεση αυτή αναφερόταν στις έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ ουσιαστικά μιλάμε για μία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είναι το Στρασβούργο. Επίσης, ε, δεν είμαστε υπέρ του να γίνονται αναφορές ή να χρησιμοποιούνται αναφορές ή πρωτοβουλία των πολιτών προκειμένου να παρακαμφθούν οι συνθήκες ή ε, η κείμενη νομοθεσία η οποία υφίσταται, όπου θα πρέπει να ζητά περισσότερο μία νομική γνωμοδότηση και επίση, για όλους αυτούς τους λόγους ήμασταν κατά της έκθεσης αυτής. Αφού όμως η έκθεση αυτή πρέπει να δει το φως ημέρας, παίξαμε και εμείς το παιχνίδι, καταθέσαμε τροπολογίες, πολλές όντως, με πολλούς υπογράφοντες, στις οποίες προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να επανέλθουμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Γιατί άκουσα τον κύριο Τσίτζεστερ αλλά και εμεί στη Γαλλία κάνουμε την αυτοκρατική μα. Γνωρίζουμε ποια είναι τα προνόμια και ποια τα μενεκτήματα από τη χρησιμοποίηση του Στρασβούργου. Σαφώ υπάρχει ένα σημαντικότατο περιθώριο βελτίωση, αλλά και κάποια σημεία δεν συμφωνούμε καθόλου. Μέσω τροπολογιών προσπαθήσαμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αυστηρότητα σε κάποια πράγματα, να γίνεται αναφορά των πραγματικών αριθμητικών δεδομένων όσον αφορά το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστο του Στρασβούργου αριθμητικά δεδομένα τα οποία κατέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμω και τα οποία θα πρέπει να ζητάμε αορίστως δεξιά και αριστερά. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στην οποία αναφερθήκαμε, μάλλον την αναφορά, ουσιαστικά γίνεται μία μόνο αναφορά αυτή τη στιγμή η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή Μόνο μία αναφορά η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή, καμία άλλη αναφορά δεν αναφέρεται, δεν πληρεί τα κριτήρια του άρθρου 191 παράγραφος 2. Μία μόνο αναφορά πληρεί όλα τα κριτήρια, δεν πρόκειται για Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών όπως υπόθηκε, αλλά για μεμονωμένη αναφορά μιλάμε. Αυτό ήθελα να αποσαφηνίσω και απευθυνόμενο στον κύριο Τσίζεστερ, ήθελα να του πω ότι ελπίζω στα συμπεράσματά του να καταγράψει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προσπαθήσαμε να επιφέρουμε μέσω τροπολογιών για την έκθεσή του. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω πολύ τον συνάδελφο Τσίτσεστερ για την έκθεσή του και να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπουλόν και την αναφέρουσα Χαίρομαι που οι αναφέροντες είναι εδώ. Εκπλήσωμαι λίγο που βλέπω στην Επιτροπή Αναφορών ότι ε, θεωρείται μη θεμητή μια αναφορά, γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν, αποφασίστηκε στην Επιτροπή αυτό που λέτε, ότι δεν ήταν παραδεκτή η αναφορά. Και είναι περίεργο να αγνοούμε τη θέληση πολιτών που είναι περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια η παράδοση της Επιτροπής είναι διαφορετική. Τέλος πάντων, δεν θα διαπληκτιστούμε εδώ κυρία Μπουλά. Και... Εγώ ως εισηγητή στην αρμόδια επί της Επιτροπή και ως μέλος και εδώ στην Επιτροπή Αναφορών θα ήθελα να πω πού αποσκοπεί η έκθεση, να διευκρινίσω και κάποια θέματα γιατί αναφέρθηκε ότι πήγαμε να την εμποδίσουμε. Στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων όλες οι ομάδες ενέκριναν την έκθεση και το γεγονός ότι θα γινόταν η έκθεση αυτή πριν από περίπου ένα χρόνο ζητήθηκε να γίνει η έκθεση και είχε μπλοκαριστεί γιατί υπήρχαν αντιδράσεις στο Κοινοβούλιο για πολύ καιρό. Εμείς θέλαμε μια έκθεση για την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά από πολλούς διαπληκτισμούς βρήκαμε το συμβιβασμό που ήταν να αλλάξει ο τίτλος και να έχουμε μία έκθεση για τις έδρες ε, του θεσμικού οργάνου και όλοι οι συνάδελφοι συμφώνησαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τελείως διαφορετικό ρόλο από τα άλλα θεσμικά όργανα στην Ένωση γιατί είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο από τους ε, πολίτες με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, είναι ισοδύναμο ε, ως νομοθέτης με το Συμβούλιο και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από τα άλλα όργανα. Γι' αυτό η Επιτροπή η συνταγματική θεωρεί ότι για τη ρύθμιση της έδρας, του χρονοδιαγράμματος εργασιών, τον, τον τρόπο εργασίας του Κοινοβουλίου στο μέλλον θα πρέπει να ισχύουν άλλοι κανόνες από ότι για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και τις αρχές που προφανώς ε, αποφασίζονται και μαζί με τα κράτη-μέλη, ανάλογα με την έδρα τους. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το θέμα έχει όπως το έθεσε ο κύριος Τσίτσεστερ από τότε που ε, δημιουργήθηκε δεν ήταν, ήταν μια συνέλευση, όχι άρμεσα εκλεγμένη, ε, δεν ήταν ε, νομοθετικό όργανο και είχαν πει ότι θα συναντούν στο Στρασβούργο γιατί εκεί ήταν και το Συμβούλιο της Ευρώπης που είχε συνέλευση και από το 58 είχε πει το Κοινοβούλιο ότι εμείς θέλουμε να είμαστε στην ίδια πόλη που βρίσκεται το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πρέπει να γίνονται διαπραγματεύσεις συνεχής μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων αυτών. Δεν μπορεί να είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Από τότε και μέχρι σήμερα το Κοινοβούλιο πάντοτε ήθελε διακοπή από την Πρόεδρο. Πρέπει να σας διακόψω γιατί πέρασε η ώρα. Καλώς. Με συγχωρείτε. Συντομεύω λοιπόν. Να πω ότι θεωρώ ότι είναι καλή η γνωμοδότηση του συναδέλφου Τσίτσεστερ. Εκπλήσωμαι ε, κάπως διότι έχουμε τώρα μια πίστευτη πληθώρα τροπολογιών από τους Γάλλους συναδέλφους και θα πω μόνο το εξής πάνω σε αυτό. Εδώ πρόκειται για την αυτοκατανόηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν θέλετε. Δηλαδή, αν εμείς ε, αντιλαμβανόμεθα τον εαυτό μας ως εκπροσώπων των πολιτών ε, σε, στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα θεσμικά όργανα και θα αποφασίσουμε οι ίδιοι πώς θα δουλεύουμε, πού θα δουλεύουμε κλπ. Δεν είναι εθνικό το θέμα και απογοητεύομαι λίγο διότι κάποια μέλη του Κοινοβουλίου το κάνουν το θέμα εθνικό. Όλους μας θίγει. Είμαστε ευρωβουλευτές και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θίγονται ανεξάρτητα από την ε, ε ηθαγένεια. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι ε, μια χώρα όμοιρος των άλλων εδώ. Ε, είναι θέμα συνταγματικό. Τελευταία λέξη. Σε αντίθεση με τις μέχρι τούδε αποφάσεις του Κοινοβουλίου δεν πρέπει πάλι να κάνουμε προσπάθεια επί της ουσίας να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να ανοίξει ο δρόμος, να αποκτήσει το Κοινοβούλιο το δικαίωμα να αλλάξει το θέμα αυτό, να το αποφασίσει μέσα από τροποποίηση το, της συνθήκης. Και καλό θα ήταν να αποφανθεί ε, προς αυτή την κατεύθυνση και η Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βαλέσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την πλήρη μου στήριξη στον κύριο Τσίτσεστερ υπέγραψα την ε, αναφορά αυτή με όλη μου την καρδιά. Την πιστεύω ακραδάντως. Νομίζω ότι συλλογικά χτυπάμε το κεφάλι μας όλοι σε αυτό τον ε, τοίχο. Όσο οι πολιτικοί ηγέτες της χώρες μας νύπτουν τα σχήρας μας, τα σχήρας τους, εμείς δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Δεν θα πρέπει να το συζητούμε τότε. Όχι. Καλώς το συζητούμε. Μέχρι ότου να βρεθεί μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα αυτό, με ικανοποιητική σχέση κόστους-οφέλειας. Έχουμε 164 ε, τροπολογίες. Πολλές από αυτές θέλουν τελικά οι προσπάθειές μας να εκτροχιαστούν. Καλό θα ήταν να έχουμε μία απλή και συγκεκριμένη γνωμοδότηση για να ξέρουμε όλοι τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Θα σας στηρίξω μέχρι τέλους. Ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν παρακαλώ. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Χαίρομαι γιατί είναι ευρία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο η άποψη ότι βεβαίως και έχουμε το δικαίωμα να το συζητούμε. Ο το έβαλε στις όχι ο Θεός ο ίδιος. Μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι δεν απέχει και πολύ από το Θεό, αλλά εν πάση δεν είναι. Μετά το δημοψήφισμα στη Γαλλία, το 1992, ο Μιτεράν το έβαλε αυτό στη συνθήκη, όπου το ναι ήταν πολύ ισχνό. Το 1992 και μετά το δανέζικο όχι, συγγνώμη που εμείς πρώτα σας βαρύναμε, εμείς είχαμε ένα πολύ διακριτικό όχι στη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά έγινε δημοψήφισμα στη Γαλλία διότι δήλωσε ο, Μαριά, Μιτεράν ότι η Μαριάν είναι υπέρα. Εμείς ως Δανείοι πετύχαμε το opt-out, το οποίο βαραίνει εμάς ως Δανούς, όχι το υπόλοιπο Κοινοβούλιο και όχι την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Συμφωνία του Ενδιβούργου, ο Μιτεράν επέβαλε 12 ολομέλειες να πάνε στο Στρασβούργο και μπήκε για πρώτη φορά μετά αυτό στη συνθήκη του Άμστερνταμ. Μόνο αν συγκρίνεται το Μιτεράν με το Θεό, που δεν νομίζω ότι κάνει κανείς από εσά εδώ, ε, δεν θα συζητείτε το θέμα αυτό. Ιδαλλιώ βεβαίω έχουμε και το δικαίωμα να το συζητούμε για να μην σα πω ότι μπορεί να έχουμε και το δικαίωμα να το αλλάξουμε κιόλα. Ευχαριστώ. Να ολοκληρωθεί παρακαλώ η συζήτηση. Την γνωμοδότησα την ψηφίσουμε στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να βρεθεί συνένεση για τις συμβαστικές τροπολογίες με τον κύριο Τσίτσεστερ. Πράγματι, θα επιδιώξω να έχουμε αντάντα, Συμφωνία κυρίων. Ευχαριστώ. Τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει χρόνος και δεν είναι και εδώ κιόλας ο κύριος Μακμίλαν Σκότ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, γιατί ο χρόνος τρέχει. Να ενημερώσω του συναδέλφους ότι 11 Ιουλίου είναι η καταληκτική προθεσμή για τις τροπολογίες. 11 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα. Η κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Μακμίλαν Σκότ δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει σήμερα και μου ζήτησε να διαβάσω την παρουσίαση που θα έκανε για την έκθεσή του, αν μου το επιτρέπετε, ή τέλος πάντων τι θα κάνουμε τώρα. Δώστε μας την παρουσίαση για να τη βάλουμε στα πρακτικά. Εντάξει, αν είναι αυτό μέσα στο ε, πλαίσιο των κανόνων μας... Μπορείτε, προβλέπετε. Δώστε μας ε, γραπτός την ε, παρουσίαση. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ίδιο ισχύει για τη συνάδελφο Μπασέσκου η οποία πρόκειται να γεννήσει σύντομα και δεν μπορεί να έρθει. Έχω τις παρατηρήσεις της, θα την εκπροσωπούσα, θα την παρουσίαζα εγώ αντί για εκείνη, θα τις δώσω στα πρακτικά να συμπεριληφθούν. Ευχαριστώ. για τις συνεδρίες.